Buenos días. En la... Καλημέρα σας. Ας δούμε, ε, ας ενημερώσουμε καταρχάς ε, τι έγινε στη συνάντηση των συντονιστών. Ε, υιοθετήθηκε μια απόφαση για την απαγωγή παιδιών στην Ιαπωνία. Μετά κάποια άλλα θέματα αποφασίστηκε να αναβληθούν μέχρι τον Απρίλιο, ε, ενώ άλλα θέματα θα μπουν στην ε, ε, συνεδρίαση του Μαρτίου. Οι 888, 217, 218, 219, 423, 219, η 336 2012, ε, και διάφορες άλλες αναφορές 2012 ε, παραδείγματος θα μπουν στις ε, στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Η 38-2020 θα εξεταστεί από την Επιτροπή μας όταν έχουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η 171 του 2013 περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη του Ιουνίου. Τώρα, ε, γνωμοδοτήσεις στην, ε, για την ετήσια έκθεση για την εξαγωγή όπλων στην Αφρική, για τη μείωση των ε, ανισοτήτων όσον αφορά την αμοιβή της εργασίας. Ο κύριος Φράγκος είναι ο εισηγητής από την ομάδα ECR. Θα είναι ο εισηγητής για την ε, της έκθεση για την πρόοδο με την Τουρκία του 2019 αποφασίσαμε να αναβάλουμε την επίσκεψη μας στην Πολωνία για το δεύτερο εξάμεινο για, την, ε, για το θέμα των ε, υπηρεσιών προστασίας στη Γερμανία θα ανατεθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα γίνουν δύο ακροάσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και διοργανικές ε, ε σχέσεις. Επίσης, ζητήσαμε από την υπηρεσία ε, πληροφοριών να μας δώσει κάποιες πληροφορίες και τα σημεία 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης θα ε, εξεταστούν με τη γραπτή διαδικασία ε, επίσης ε, εγκρίναμε το πρόγραμμα για την ακρόαση και σύμφωνα με το άρθρο 2.30 ε, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Πρόεδρος θα ενημερώσει τους αναφέροντες για το ECCI με μια επιστολή και στις 24 Μαρτίου του 2020 θα γίνει σχετική ακρόαση. με την βοήθεια της Επιτροπής ΑΦΚΟ ε, θα ε, εξετάσουμε τα θέματα αυτά και τώρα ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη σημείο 17 μια αναφορά ενός Γερμανού υπηκόου σχετικά με την αλλαγή του ονόματος ε, του της αίθουσας ε, ε, της Ολομέλειας ε, στις Βρυξέλλες, στο κτίριο των Βρυξελών. Έχετε πέντε λεπτά για να παρουσιάσετε το θέμα σας. Ευχαριστώ. Ε, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της Επιτροπής Αναφορών, πριν από μερικές, ε, μερικούς μήνες έγραψα ιστορία στην Ευρώπη. δεν... Ε, χρειάζεται να σα υπενθυμίσω ότι ακόμα συζητείται η πρότασή μου αυτή. Θα ήθελα όμως να σα θυμίσω τι έγινε για να βοηθήσω του μελλοντικού βιογράφου μου. Ε, Το περασμένο Νοέμβριο ε, έληξε η έξι δεκαετία του θέματος της διπλής έδρας του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να σας πω πώς βρήκα ένα παραθυράκι στη, στη διάταξη της ε, ε, συνθήκης που ορίζει την έδρα του Κοινοβουλίου. Λέει ε, η διάταξη αυτή το, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στο Στρασβούργο 12 φορές το χρόνο. Δεν λέει ποιο Στρασβούργο όμως. Οι περισσότεροι βεβαίως ε, υποθέτουν το Στρασβούργο της Γαλλίας, 450 χιλιόμετρα από εδώ. Αλλά αυτό γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική λύση μέχρι τότε. Τώρα υπάρχει Στρασβούργο ε, Βρυξέλλες, Στρασβούργο Βρυξελών, 400 μέτρα απόσταση από εδώ. Αν το ημικύκλιο ονομαστεί Στρασβούργο, μπορείτε να συνεδριάζετε εκεί κάθε μήνα χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε ούτε μία λέξη μέσα στις συνθήκες. Γιατί αυτό ήταν απαραίτητο διότι η δεύτερη έδρα είναι μια σπατάλη χρημάτων. Ε, ανανομοθετική περίοδο κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ. Επίση είναι χάσιμο χρόνο. 100 ώρες ε, το χρόνο χάνετε όλοι σα για τα ταξίδια μπρο πίσω στο Στρασβούργο. Και είναι και σπατάλη ε, χώρου. Τα γιγαντιαία κτίρια του Στρασβούργου είναι άδεια 300 μέρες το χρόνο. Ε, φαντάζεστε πόσο πιο χρήσιμα θα ήταν αν χρησιμοποιούνταν για κάτι που πραγματικά έχει ανάγκη η Ευρώπη. κάτι που, ε, παραδείγματο χάρη, ένα πανεπιστήμιο ε, για όλους αυτούς που δεν μπορούν να βρουν ε, δουλειά στην Ευρώπη ή ένα πολυτελές καταφύγιο ε, για πρόσφυγες. Αλλά το πιο σημαντικό, η δεύτερη έδρα είναι μια σπατάλη για τη γη. Κάθε μέρα, κάθε, κάθε χρόνο παράγεται εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα έχετε κηρύξει έκτακτη ανάγκη για το περιβάλλον. Ε, ορίστε, η απόδειξη του τι έκανα στην αίθουσα του, της Ολομέλειας. Ζητώ λοιπόν από το Κοινοβουλίο να δώσει την γραφειοκρατική του ευλογία ε, στην αλλαγή αυτού του ονόματος που σας προτείνω. Εδώ έχω ετοιμάσει και την πινακίδα. Απλώς το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώσει ε, την απόφαση αυτή και είμαι έτοιμος να καρφώσω την πινακίδα. Οι διαχειριστές του κτηρίου θα πρέπει να με αφήσουν να ε, βάλω την πινακίδα αυτή στον τοίχο. Κάποιοι θα πούν ότι όλα αυτά είναι ένα ανέκδοτο και συμφωνώ πραγματικά αυτά τα πήγαινε μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου είναι κάτι το χαοτικό. Αλλά μερικές φορές πρέπει να σας πω, σχετικά με τα ανέκδοτα, ότι αν επί 60 χρόνια ε, συνεχίζετε να λέτε το ίδιο ανέκδοτο, δεν είναι πια αστείο. Σας παρακαλώ λοιπόν να υποστηρίξετε την αναφορά μου. Είναι η, η ευκαιρία σας να αλλάξετε κυριολεκτικά το μέλλον της Ευρώπης. Ας μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το θέμα. και εύχομαι αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΤΗ να είναι η ιστορική στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτέλους θα σταθεί στο ύψος του και θα αναλάβει τον έλεγχο της μοίρα του, του πεπρωμένου του. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν. Κυρία Κρίστενσεν, καλημέρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θυμίζω ότι το ζήτημα της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ρυθμίζεται στο πρωτόκολλο 6 σχετικά με την, τον τόπο το, της έδρας των θεσμικών οργάνων και των διαφόρων οργανισμών της Ένωσης. Εις ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πρωτόκολλο προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο θα έχει την έδρα του στο Στρασβούργο ε, όπου οι 12 σύνοδοι συν την ε, σύνοδο για τον προϋπολογισμό θα λαμβάνουν χώρα. Οι πρόσθετες ε, σύνοδοι της Ολομέλειας θα λαμβάνουν χώρα στο, στις Βρυξέλλες. Το πρωτόκολλο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των συνθήκων και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με, στα πλαίσια αναθεώρησης συνθήκων. Η Κομισιόν θεωρεί αδιαμφισβήτητο ότι η αναφορά στο πρωτόκολλο υπαριθμών 6 στο Στρασβούργο ως το χώρο όπου θα διεξάγονται οι Ολομέλειες νομικά αναφέρεται στη γαλλική πόλη του Στρασβούργου, στην περιοχή της Αλσατίας και όχι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή τόπο που να ονομάζεται Στρασβούργο. Γι' αυτό νομικά δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί η λέξη Στρασβούργο στο πρωτόκολλο με τρόπο τέτοιο ώστε να συνάδει με την πρόταση να γίνονται οι 12 ολομέλειες στην ε, αίθουσα της Ολομέλειας των Βρυξελών εάν με ονομαζόταν σε αίθουσα Στρασβούργο. Ευχαριστώ. κύριος Αλιμόφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα αντικαθιστώ τον συνάδελφο Ράντεφ που ζητεί συγνώμη για την απουσία του. Και θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση μας. Τη θέση της πολιτικής μας ομάδας. Όπως αναφέρει ο αναφέρον, έχουν γίνει συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το ενδεχόμενο μιας έδρας και υπήρξαν και αναφορές σχετικές. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Από τη μία έχουμε τις συνθήκες και οι αποφάσεις για την τροποποίηση των συνθήκων μπορούν να ληφθούν μόνο από τα κράτη-μέλη. Όμως, πολύ συχνά ακούμε ευνοϊκές συνέπειες επιπτώσεις για μια τέτοια τροποποίηση της συνθήκης. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι το Κοινοβούλιο είναι διαιρεμένο σε αυτό το θέμα. Εξ του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι το καλύτερο θα ήταν αν η Επιτροπή λάβει απόφαση αφού ακούσει όλες τις γνώμες και μετά θα αποφανθεί επί της ίδιας της αναφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φίρς. Ε, βρίσκομαι εδώ όχι για το θέμα του single seat που μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να πω ότι αναφορά που σε γίνεται σήμερα έχει πολύ ε, ε, περίεργη μορφή. Ε, μιλάει για βάφτιση μιας ε, αίθουσας. Καταλαβαίνω βέβαια το, τα επιχειρήματα του συναδέλφου, γιατί έχουμε τόσο καιρό που ακούμε σοβαρά επιχειρήματα για αυτό το θέμα. Ξέρουμε βέβαια ότι οι συνθήκες δεν ε, μας δίνουν πολλά δικαιώματα σε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι μία από τους πρώτους ευρωβουλευτές. Ήμασταν πέντε το 2006, η κυρία Μάλστρομ, που μαζέψαμε τρία εκατομμύρια και υπογραφές και τις ε, υποβάλαμε στην Κομισιόν ε, εκείνη την εποχή ζητώντας ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο όμως επιμένει στην ε, θέση αυτή. Από ό,τι θυμάμαι, ε, έφερε το Κοινοβούλιο ε, το θέμα αυτό στο, στη Σύνοδο του Συμβουλίου. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον Πρόεδρό μας να εκφράσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εντωμεταξύ από ψηφοφορία σε ψηφοφορία, όποιο και αν είναι το θέμα, παραδείγματο χάρη για το Green Deal, για τι κλιματικέ αλλαγέ, 450 βουλευτέ ψήφισαν υπέρ και για την έκθεση αυτή. Και είναι οι ίδιοι 400-500 συνάδελφοι κάθε φορά που τάσσονται υπέρ της ε, ενιαίας έδρας. Αναφέρομαι τώρα στο σημείο 7. Δεν είμαι ε, αντίθετη στο να έχουμε ένα καταφύγιο για τους άστεγους, εντάξει, αλλά εμεί κάναμε προτάσεις πιο ακαδημαϊκές. Παραδείγματο χάρη είναι να γίνει πανεπιστήμιο στην έδρα του Στρασβούργου. Τα πράγματα μπλοκάρονται όμως στο Συμβούλιο. Ε, σκεφτείτε τι έγινε όταν έπρεπε να αλλάξουν έδρα οι δύο οργανισμοί που βρίσκονταν στην, ε, στο Ενωμένο Βασίλειο, ιδίω ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η πρόταση για το Στρασβούργο τότε ήταν ιδανική. Πραγματικά όλες οι συνθήκες ε, υπήρχαν, αλλά ε, δεν ε, άλλαξαν οι θέσεις. Και για πρώτη φορά πρέπει να σας πω ότι ε, ακούστηκαν κάποιοι τρίγμοι από το περιβάλλον της Άγγελας Μέρκελ, που μέχρι τότε δεν ήθελε να αλλάξει στάση για το θέμα αυτό και πραγματικά και εκείνη πρότεινε ε, το Στρασβούργο ως μελλοντική έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα φάρμακα που τελικά βέβαια ξέρουμε ότι ε, την κέρδισε το Άμστερνταμ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, ε, όπως και πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές, Ε, είμαστε ε, υπέρ του να μην αμφισβητήσουμε ε, το θέμα της έδρας πλέον. Το θέμα αυτό το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ διάφορες λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη που και από την άλλη μεριά αναφερόμαστε πάντα στις διατάξεις της συνθήκης, ε, πρέπει να βρούμε μία λύση που να είναι επωφελής για όλους. Αλλά αυτό ε, που είναι ε, πραγματικά ανυπόφορο είναι να μας μπλοκάρει το Συμβούλιο. Φυσικά η αναφορά αυτή είναι διατυπωμένη με έναν τρόπο όχι και τόσο ακαδημαϊκό, για να το πω έτσι ευγενικά, αλλά ε, επί της ουσίας είναι, αναφέρεται σε ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολεί εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο αναφέρον θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη προτείνει την αλλαγή του ονόματος της αίθουσα της Ολομέλειας εδώ στις Βρυξέλλες και να την ονομάσουμε Στρασμπουργκ. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Αυτό το πρόβλημα συζητείται χρόνια στο Κοινοβούλιο. Είναι θέμα ιστορικό, ακόμα και κατά την ε, ε, διατύπωση των ε, των ε, συνθήκων, οι Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο αναφέρθηκαν. Πάντως πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση. Αφού μιλάμε για την ανάγκη μείωση των εκπομπών. Εξαιτίας αυτού του ιστορικού στοιχείου, αυτού του δεδομένου, ότι κάθε μήνα πρέπει να μετακινούμε όλες τις υπηρεσίες από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, δεν νομίζω ότι δίνουμε καλό παράδειγμα στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Κάθε φορά που πηγαίνω ερχόμαστε, κάθε μήνα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες συζητήσεις με θέμα τη μία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί πραγματικά ε, διασπαθίζονται πάρα πολλοί πόροι και σε οικονομικό επίπεδο. Χρησιμοποιούμε τα χρήματα των πολιτών και δεν πρέπει να τα σπαταλούμε πηγαίνοντας από και προς προς το Στρασβούργο. Το Κοινοβούλιο έχει περάσει έναν αριθμό ψηφισμάτων. Αναφέρω ιδιαίτερα αυτό στις 16 Φεβρουαρίου του 2017, όπου ζητείται η αλλαγή, τροποποίηση στις συνθήκες και η ανάγκη για λήψη της σχετικής απόφασης. Όπως είπα, δεν είμαι ευτυχής με τη διατύπωση της αναφοράς αυτής, ούτε πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση αλλάζοντα το όνομα της αίθουσα της Ολομέλειας. Όμως μπορώ να καταλάβω την ουσία της αναφοράς και πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα για να ληφθεί μια απόφαση. Είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς την συγκεκριμένη αναφορά, όπως σας είπα. Δεν νομίζω ότι έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Λόκα. Ευχαριστώ, η κυρία Στανόκα. Ε, υποστηρίζω ότι πρέπει να είναι παραδεκτή, να ενημερωθεί και ο αναφέρον, ο οποίος σίγουρα θα γνωρίζει τα πολλά ψηφίσματα σχετικά του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να προωθήσουμε την αναφορά αυτή στην ΑΦΚΟ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήματα. Θέλω μόνο να θυμίσω στον κύριο Σέμσροτ ότι δεν έχει εκείνος την ευρεσιτεχνία για αυτό το θέμα. Παλιότερα, το 2008, όταν ε, έπαθε ζημιά η οροφή, ένα κομμάτι της οροφής ε, της αίθουσας της Ολομέλειας στο Στρασβούργο ε, έπαθε ζημιά. Κανείς δεν ήταν ευτυχώς στο αίθουσα εκείνη την ώρα και δύο, δύο ολομέλειες έγιναν στις Βρυξέλλες. Δεν πήγαμε στο Στρασβούργο. και ο συνάδελφός μου Άλαν Σμιθ ε, που ήταν από τη Σκοτία Ευρωβουλευτής, τώρα είναι Εθνικός Βουλευτής στη Βουλή των Κοινοτήτων, είχε εκφράσει αυτή την ιδέα και την κυκλοφόρησε και είχε πει ακριβώς να ονομαστεί Στρασβούργο η αίθουσα της Ολομέλειας εδώ. Οπότε δεν είστε εσείς ο πατήρ της ιδέας. Ε, ε, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν είστε ο πρώτος που είχε αυτή την ιδέα, η οποία όμως είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Άουκεν. Συγγνώμη που άργησα και έχασα τη συζήτηση θυμίζω κάτι πολύ σημαντικό σε όλους. Το Στρασβούργο δε, το, το 98 με τη συνθήκη του Άμστερνταμ μπήκε στις συνθήκες στο Στρασβούργο. Ε, ε, υπήρχαν λόγοι, είτε το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι εκεί και όχι, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν εκεί, χρησιμοποίησε τις εγκαταστάσεις και μετά ε, έπρεπε να έχει δικό του χώρο το κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στις... Στην Ισπανία δεν μπορεί να είναι το κοινοβούλιο μακριά από το κέντρο εξουσίας, να πάει στη Βαλένσια, πρέπει να είναι στο κέντρο εξουσίας. Και γι' αυτό τότε ε, είχαμε τη συνθήκη του Μάστερ και ο Μιτερό είχε πει ε, ότι θα έκανε δημοψήφισμα στη Γαλλία, έγινε και τα αποτελέσματα δεν ε, ήταν ε, υπέρ του. Εμείς είδαμε τη Γαλλία να επιμένει να συμπεριληφθεί στη συνθήκη η υπόθεση των 12 ολομελιών στο Στρασβούργο. Αλλά πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει σχετικά με τα θέματα που το αφορούν. Και έχουμε τώρα αυτή την κατασπατάληση χρήματος. Το Στρασβούργο είναι πολύ καλό. Έχουμε το, στο Στρασβούργο είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, είναι καλό το Στρασβούργο, αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί και εμείς έχουμε εξουσία. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Ζέμσρωτ, για να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επί της ουσίας. Απλώς έχουμε διαφορετική άποψη για το ποια είναι η καλύτερη μέθοδος και αν δούμε τα προηγούμενα ε, χρόνια ε, θα καταλήξουμε ότι η καλύτερη και τελευταία επιλογή είναι να αλλάξουμε το όνομα της αίθουσας της Ολομέλειας. Συμφωνώ και με την κυρία Ρής και με την κυρία Άουκεν και την αντιπρόεδρο, την κυρία Σδανόκα. Δεν ε, διεκδικώ την ιδέα ως δική μου, αλλά ε, μπορούμε σε θεσμικό επίπεδο όλοι να μοιραστούμε την ιδέα. Ευχαριστώ και για την, την Κομισιόν για την απάντηση. Μπορείτε να μου δώσετε αποδείξεις ότι πρόκειται για το Στρασβούργο στη Γαλλία, γιατί εγώ δεν το βρήκα αυτό που λέτε στις συνθήκες. Βέβαια, δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί ένα ε, εργαλείο, μια μεθοδολογία θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Ένβη Αναφορά για να μας αναφερθεί στα περιβαλλοντικά ωφέλη που θα επιφέρει η αλλαγή του ονόματος και την Επιτροπή Προϋπολογισμού γιατί θα έχουμε εξοικονομήσει στην Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί θα έχουμε ένα ε, πανεπιστήμιο για ανθρώπους που απέτυχαν παλιότερα και άλλες επιτροπές. Και αφού όλες οι αυτές οι επιτροπές θα αποφανθούν, θα θέσουμε ψήφισμα ε, στην Ολομέλεια προς ψήφιση ούτως ώστε επισήμως το ημικύκλιο στις Βρυξέλλες να ονομαστεί Στρασβούργ. Και μπορούμε και το ημικύκλιο του Στρασβούργου να το ονομάσουμε Βρυξέλλες έτσι για να υπάρχει ισορροπία και να πηγαίνουμε εκεί για την ε, συζήτηση για τον προϋπολογισμό, την Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακούσαμε τον αναφέροντα, ακούσαμε την Κομισιόν, ακούσαμε τα μέλη της Επιτροπής και τώρα θα, η πρόταση είναι να μείνει ανοιχτή η αναφορά όπως αναφέρθηκε και πριν. Εμείς όταν τη, λάβαμε, τη στείλαμε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και θα περιμένουμε τη γνωμοδότηση από εκεί και Ήδη το Φεβρουάριο του 2017 το Κοινοβούλιο εδήλωσε ότι είναι υπέρ μιας και μόνης έδρας. Ε, έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 18, είναι η αναφορά 1140 του 2018 από το Φερνάντο Νοβέγια εξ ονόματος μιας ε, ισπανικής οργάνωσης ε, που καταπολεμεί τον αμίαντο. Δεν είναι δεν είναι εδώ αναφέρον, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Βίλιαμ Τάιλερ από την Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Έχετε λάβει ήδη τις παρατηρήσεις μας. Ε, θα σας αναφέρω μόνο τα κυριότερα στοιχεία και τις τελευταίες εξελίξεις, τις πιο πρόσφατες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απολύτως ότι ο αμύαντος είναι αντικείμενο μεγάλης ε, ανησυχίας και απαιτεί ε, τα κατάλληλα μέτρα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των κρατών μελών. Και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό και εκτιμένο για τον αμίαντο. Ένα παράδειγμα μόνο στα θέματα ε, των επαγγελματικών ασθενειών έχουμε μια οδηγία που είναι ειδικά ε, αφιερωμένη στην έκθεση στον αμίαντο. Είναι η οδηγία 2009-148, η λεγόμενη και οδηγία ε, για τον αμίαντο. Λοιπόν, ε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σωστά επιτόπου σε κάθε κράτος μέλος. Και γι' αυτό θέλουμε να τονίσουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που ε, έχουν εδώ τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι για να υποστηρίξουμε αυτά τα πολύ σημαντικά τους καθήκοντα, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε έναν οδηγό με τις βέλτιστες πρακτικές για τον αμύαντο, για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, αλλά και τους επιθεωρητές εργασίας, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά. Δεύτερον, και το αναφέρουμε αυτό στις παρατηρήσεις μας, μία απόφαση για την απομάκρυση του αμοιάντου από κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά εξαρτάται από ε, παράγοντες και παραμέτρους ε, που αφορούν ειδικά το κάθε κτίριο. Και αυτή την απόφαση ε, τα κράτη-μέλη ε, μπορούν μόνο να την πάρουν, γιατί αυτά είναι καλύτερα σε θέση να καταλάβουν, να αποφασίσουν αν το, η απομάκρυνση του αμοιάντου από ένα κτίριο είναι το πιο σωστό και κατάλληλο μέτρο. Μετά, πρέπει να αναφερθώ σε μία σύσταση της Κομισιόν για το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, για τις επαγγελματικές νόσους και ιδιαίτερα το άρθρο 2 που λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα ε, για να ορίσουν τα κριτήρια μέσω των οποίων αναγνωρίζονται οι επαγγελματικές νόσοι μεταξύ των οποίων και αυτές που σχετίζονται με την έκθεση στον αμίαντο. Και να αναφερθώ εν συντομία στα συμπεράσματα των παρατηρήσεών μας. Εκεί λέει ότι όσον αφορά την ασφάλεια και η υγιεινή στην εργασία όλα τα θέματα που ο αναφέρον θέτει υπόψη αυτή της επιτροπή υπάγονται στι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Άρα η Κομισιόν έχει την άποψη ότι θα πρέπει να τα αναλάβουν τα θέματα αυτά και να τα αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Και τέλος, επιπλέον αυτών θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κομισιόν πρόσφατα... Ε, ανέθεσε στην ΕΚΑ, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για, για τα Χημικά Προϊόντα, που βρίσκεται, έχει έδρα στη Φιλανδία, ανέθεσε λοιπόν στον ΕΚΑ να πραγματοποιήσει μία μελέτη ε, που να ε, εξετάζει ε, την αποτελεσματικότητα των ορίων σχετικά με τον αμίαντο που θέτει η σχετική οδηγία και την καταλληλότητα των ορίων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Σαλίβα. Ευχαριστώ. Ο αμίαντος είναι από τα υλικά που αποδεδειγμένα μπορεί να προκαλέσουν ίνωση και καρκίνο. Πρέπει λοιπόν να απομακρυνθεί το ταχύτερο δυνατόν από όλα τα δημόσια κτίρια και όταν βλέπουμε τέτοιες αναφορές όπου έχουμε ε, δημόσια κτίρια ή σταθμούς του μετρό στην, υπάρχουν στην Ισπανία με αμίαντο σταθμή. Είναι πολύ ανησυχητικό. Σε εθνικό επίπεδο αποφασίστηκε ότι πρέπει σταδιακά να απομακρυνθεί ο αμίαντος από όλα τα δημόσια κτίρια. Υπήρχε και ε, ψήφισμα του Κοινοβουλίου από το 2013 και τώρα μπορούμε να πούμε ότι ε, έχουν περάσει και 19 χρόνια από τη Συμφωνία του 2001. Ε, είχαμε χρόνο να απομακρύνουμε τον επικίνδυνο αμίαντο, επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στις ισπανικές αρχές ώστε να αποφύγουμε έναν πραγματικό κίνδυνο για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Δεν είναι εδώ αναφέρον. Η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή ε, πάνω στη βάση των όσων είπε ο κύριος Σαλίμπα και θα δούμε τι μέτρα θα λάβει η Κομισιόν στο μέλλον για τον αμίαντο. Πάμε παρακάτω. Έχουμε την 171-2019 ε, από Γερμανό σχετικά με την θνησιμότητα των εντόμων λόγω του φωτισμού των δρόμων. Δεν είναι αναφέρον εδώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοβάσεβιτς από την ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην παρατήρησή μας πρόσφατα που σας τη δείξαμε δεχόμαστε ότι ο τεχνητή το φωτισμός είναι κίνδυνος για τους επικονιαστές και τα, κυρίως τα νυχτερινά, νυχτόβια έντομα που ε, δραστηριοποιούνται το βράδυ. Τονίσαμε επίσης ότι ενώ το πρόβλημα εμένει, σε ενωσιακό επίπεδο δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το φωτισμό των οδών, ε, αυτό είναι πρωταρχικά αρμοδιότητα των κρατών μελών είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να κάνει σε ενωσιακό επίπεδο η Κομισιόν να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη, τις αρχές των κρατών μελών, και να για να προωθήσουν ε, πιο φιλικές τεχνολογίες, πιο φιλικό φωτισμό των δρόμων με προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουμε αρμοδιότητα ρυθμιστική. Θυμίζω επίσης ότι ο κανονισμός Eco Design οικολογικού σχεδιασμού δεν ε, εμποδίζει την εμπορία και άλλων τεχνολογιών, αλλά ο κανονισμός eco-design δεν μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένους τύπους τεχνολογίας. Αναγνωρίζουμε λοιπόν μεν το πρόβλημα, πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι οι δράσεις προαιρετικές. Και εις ό,τι αφορά την αρμοδιότητα, παραπέμπουμε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Σαλίμπα. Ευχαριστώ τον αναφέροντα τη απουσία του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αναφορά, ιδιαίτερα όταν ε, έχουμε υπόψη μας τους επικονιαστές που οι αριθμοί τους μειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι μεγάλο τώρα, γιατί οι επικονιαστές είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματός μας και τους χρειαζόμαστε για να έχουμε ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Σημειώνω αυτό που είπε η Κομισιόν, ότι δεν υπάρχει ε, ενωσιακή αρμοδιότητα ε, για κανονισμούς σε αυτό το θέμα, αλλά καλό την Κομισιόν να προσπαθήσει και να ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση της ανάληψης δράσης σχετικά, γιατί αν όλοι κάνουν αυτό που πρέπει, αν όλοι κάνουν μια μικρή προσπάθεια και αν έχουμε σωστή καθοδήγηση ε, με κανονισμό από την Κομισιόν θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Σίγουρα πρέπει να αναλάβουμε δράση και γι' αυτό η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να σταλεί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, στην Επιτροπή ΕΝΒΗ, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ούτω ώστε να γνωμοδοτήσουν και εκείνοι. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση και να ευαισθητοποιούμε την Κομισιόν ώστε αυτή να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και τον κύριο Σαλίμπα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή. Θα την στείλουμε και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Αλλά επίσης θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, συντάξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ε, σωστή χρήση του φωτισμού ώστε να ε, προκαλεί λιγότερες, ε, ζημιά, λιγότερες βλάβες στα έντομα. Φυσικά δεν μπορεί να νομοθετήσει σχετικά η Κομισιόν, αλλά ίσως οι κατευθύνες γραμμές θα ήταν χρήσιμες για τις τοπικές αρχές. Ωραία, περνάμε στο σημείο 20 της ημερίας διάταξης, αναφορά 1694 του 2014, που υποβλήθηκε από τον Ζωακίν Πέρες Κόμες από την Ισπανία σχετικά, ε, μάλλον από εκ μέρους της οργάνωσης οικολογίστας εν Action, ε, σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης ε, της διαχείρισης των υδάτων στην Μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελόνης. Θα σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά και μετά θα έχουν δύο λεπτά οι υπόλοιποι ομιλητές να πάρουν το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. που κηρύξατε αποδεκτή την αναφορά αυτή, ε, το δικαίωμα ε, στο νερό είναι ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όπως έχει ε, δεχτεί και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης ε, ε, υπάρχει ως δικαίωμα στο, στο θεμελιώδη χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε μια τέτοια πρωτοβουλία που είχε 2 εκατομμύρια υπογραφές ε, και αφορούσε την ε, συμπερίληψη του δικαιώματος στο νερό σαν ένα από τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, γιατί το νερό είναι θεμελιώδη σημασία για, για τη ζωή του ανθρώπου. Το 2010 το δικαστήριο της Βαρκελόνης αποφάσισε ότι ε, η απόφαση για, τον, για την ίδρυυση ε, της Βαρκελόνης, ε, ο τρόπος που ανατέθηκε το συμβόλαιο αυτό ε, έγινε με αθέμητο τρόπο, με άμεση ανάθεση και γι' αυτό ε, ε, δημιουργήθηκε μια ε, επιχείρηση μεικτού χαρακτήρα για την παροχή είδατο την εξυγίαση του ύδατος, διανομή, τον εφοδιασμό πόσιμου ύδατος για δύο εκατομμύρια ανθρώπους περίπου. Έγινε ο διαγωνισμός για το 80% που ήταν το μέρος του ιδιωτικού και τελικά ε, έγινε η ανάθεση αυτή εκ μέρους ε, του Δήμου της Βαρκελόνης χωρίς ε, να κηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός. Και η πρόεδρος. Θα πρέπει να μιλάτε λίγο, να διαβάζετε μάλλον λίγο πιο αργά, γιατί οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν, λέει η πρόεδρος. Τώρα, η απόφαση του 2019 του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας ε, θεώρησε ότι υπήρξε ε, ελεύθερος ανταγωνισμός και ότι μια τέτοια απόφαση ε, είναι ε, επαρκής και σωστή νομικά, βασιζόμενη σε ένα νόμο ε, της φραγκικής περίοδου που αναθέτει το, τη σύμβαση αυτή μέχρι το 2047. Εφιστούμε την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποιες πτυχές της δημιουργίας αυτής της επιχείρησης μικτού τύπου που παραβιάζει ε, διάφορες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων ε, για τα έργα του δημοσίου. Ε, πρώτα απ' όλα, μια άμεση ανάθεση χωρίς ε, κήρυξη διαγωνισμού. Είναι ε, μία πρόκληση. Η εταιρεία αυτή, ε, η ΑΚΜΑ, ε, μπαίνει μέσα σε αυτή τη σύνθεση της ε, επιχείρησης μικτού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός. Ο Δήμος της Βαρκελόνης παίρνει αυτή την απόφαση δημιουργώντας μια μονοπωλιακή κατάσταση. Ο δεύτερο ομιλητή. Η σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα συμφέροντα τη ΑΚΠΑ είναι σαφής. Αλλά επίση, ε, ήθελα να αναφέρω κάποια άλλα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι αθέμητα. Η ΑΚΠΑ έχει μια συμφωνία με την ε, ε, με το Δήμο της Βαρκελόνης να εκπαιδεύσει δικαστές. Ε, η σύνθεση του τμήματος του δικαστηρίου ε, άλλαξε τρεις φορές και κρίθηκε από ένα τμήμα άσχετο με το θέμα. Τα τοπικά μέσα ε, μάλλον ε, πρόσφατα οργανώθηκε μια εκδήλωση ε, με, όπου ήταν εκπρόσωπος και ο, συμμετείχε και ένας εκπρόσωπος της ΑΚΠΑ καθώς επίσης και οι υπουργοί της Ισπανίας που θεώρησαν ότι μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον μονοπωλιακό τρόπο. Θεωρούμε ότι παραβιάζονται οι κανόνες σχετικά με την ύπαρξη μονοπωλίων, διότι έγινε ε, αυτή η άμεση ανάθεση. Ε, συγκεντρώνεται έτσι η διαχείριση των υδάτων ε, στα χέρια ενός μόνο φορέα. Επίσης θεωρούμε ότι παραβιάζεται η αρχή της περάσπισης του γενικού συμφέροντος γιατί η διάρκεια αυτής της σύμβασης, αυτού του συμβολέου δεν είναι αιτιολογημένη, δεν δικαιολογείται τέτοια διάρκεια. Όλες αυτές οι παραβιάσεις ε, θεωρήθηκαν ε, ε, νόμιμες όμως από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και γι' αυτό ακριβώς ε, απευθυνόμαστε στην Επιτροπή σας. Και θα θέλαμε και η Επιτροπή, του Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά, η, η ΙΝΚΟ, να η ΙΜΚΟ να εξετάσει το θέμα από την άποψη της εσωτερικής αγοράς που αφορά 3,2 περίπου εκατομμύρια κατοικούς που μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελόνης. Η Κομισιόν, η κυρία Ντίτα Κολίνσοβα. Καλημέρα. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θέλω να πω ότι το θέμα αυτό που όπως το παρουσίασαν οι αναφέροντες μέχρι πρόσφατα ήταν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο και η Κομισιόν έλαβε υπόψη την απόφαση από τον Νοέμβριο του 19 του Ανωτάτου Ισπανικού Δικαστηρίου που θεώρησε ότι βάσει ύπαρξης αποκλειστικών δικαιωμάτων ήταν δικαιολογημένη η διαδικασία που ακολούθησε η Δημόσια Αρχή και η άμεση ανάθεση θεωρείται νόμιμη από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Η Κομισιόν θα ήθελε να πει ότι για τον τομέα των υδάτων τώρα αποκλείεται ο τομέας αυτός από την οδηγία για τις παραχωρήσεις. Ούτε και παλιά ήταν αντικείμενο του παραγόγου δικαίου της Ένωσης. Αυτή ήταν η απόφαση που ελήφθη κατά τις διαπραγματεύσεις ε, για το παράγωγο δίκαιο. Ε, επίσης πάνω στη βάση προηγουμένων πρωτοβουλειών που προαναφέρθηκαν που αφορούσαν το τομέα των υδάτων και τα ύδατα καθ' αυτά. Στην ε, οδηγία για τις παραχωρήσεις, στην ιδεολογική σκέψη 40, οι παραχωρήσεις στα ύδατα συχνά είναι αντικείμενο σύνθετων ρυθμίσεων που πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα επειδή το είδωρ είναι δημόσιο αγαθό με μεγάλη αξία για όλους τους πολίτες. Ε, και μπορεί να υπάρξουν αποκλεισμοί από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για ορισμένε παραχωρήσει συμβάσεις. Και ιδίω στο παράγωγο δίκαιο, στον κανόνα για τι δημόσιε συμβάσει, υπάρχουν καμιά φορά περιπτώσει που επιτρέπουν τη χρήση διαπρα... Ε, διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη ε, υποχρέωση σε δεόντως αιτιολογημένες υποθε... περιπτώσεις, όπως αυτές που αφορούν λόγους σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, όπου η ανάθεση μπορεί να γίνει μόνο σε, συγκεκριμένο μόνο, ε, σε συγκεκριμένη μόνο επιχείρηση. Έτσι, οι νέες εξελίξεις στο δικαστικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο που εξέτασαν εκτενώς το θέμα ε, στα εθνικά δικαστήρια, η Κομισιόν δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στο θέμα που έθεσαν οι αναφέροντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τη συμβολή της στη συζήτηση. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, η εσωτερική δικαστική διαδικασία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί υπάρχει αναφορά, ε, ε, αίτηση για ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έχει υποβληθεί, οπότε περιμένουμε την τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με την αίτηση ακύρωση της απόφασης. Οι εσωτερικές δηλαδή δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ένα είναι αυτό. Να αναφέρω ακόμη ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η πρώτη σημαντική απόφαση σχετικά από το Καταλανικό Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε σαφώς ότι υπήρχαν λόγοι να πιστέψουμε ότι σε αυτή την περίπτωση και στην απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση δεν πληρούνταν και δεν έγιναν σεβαστά συγκεκριμένα άρθρα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκαιο ανταγωνισμού. Το Καταλανικό Ανώτατο Δικαστήριο είπε ότι ενδεχομένως υπάρχει καταστρατήγηση του ενωσιακού δίκαιου και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί επίση οι διαδικασίε στο ανώτατο Ισπανικό Δικαστήριο. Ε, δεδομένου αυτών των δύο πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Επίση, πιστεύω και καταλαβαίνω βέβαια αυτό που λέει η Κομισιόν ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι στην τωρινή μα ε, νομοθεσία και στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και στο δίκαιο ανταγωνισμού που επιτρέπουν απευθείας αναθέσεις μετά από διαπραγμάτευση. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, να δικαιολογούνται με κάποια βάση ορισμένων κριτηρίων και θα πρέπει να, δου, να δει η Κομισιόν αν πληρούνταν αυτά τα κριτήρια γιατί τώρα βλέπουμε ότι μια δημόσια υπηρεσία ε, ανέθεσε την παροχή ύδατος σε ένα σημαντικό κομμάτι της ε, Ισπανίας της ε, Βαρκελόνης δηλαδή, που από το 1953 δεν επέτρεπε στην εταιρεία να κάνουν αυτά που έκαναν τα τελευταία 30 χρόνια. Ε, έτοιμα προς την Κομισιόν. Επειδή η εσωτερική δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω και η ομάδα μου πιστεύει ότι υπάρχουν λόγοι ε, για τους οποίους πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα, πιστεύω λοιπόν ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Κύριο Σαλίνα. σε Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από δύο πλευρές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ε, έχει επιβεβαιωθεί προηγουμένως, έχει αναφέρει ξεκάθαρα και έχει παραθέσει και το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια έλλειψη αρμοδιότητας Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά εξαιρέσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς, όπως αυτή εδώ. Ωστόσο, η Επιτροπή, παρότι δεν είχε αυτή την ε, σαφή αρμοδιότητα, τα τελευταία χρόνια έχει συνεχίσει να ε, διεξάγει την έρευνά της. Και τώρα έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε σαφής αιτία για την αίτηση υπήρξε και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, όπου έχει αναφερθεί ότι αυτές οι υποτιθέμενες ε, παραβιάσεις ε, του, ε, του δικαίου ανταγωνισμού δεν έχουν λάβει χώρα. Γι' αυτό δεν κατανοώ γιατί πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αίτηση. Ζητώ λοιπόν να κλείσει. Ευχαριστώ. Señora Ρίβα. gracias. Señora Κυρία Ρίβα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ετούντες που είναι εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό που τους ακούσαμε σήμερα εδώ, ιδίω μετά από την απόφαση του Ανατότου Δικαστηρίου, που προτείνει τη διατήρηση του ΑΚΜΑ ως ε, ε, για τη δυνατότητα ε, ίδρυυσης της Βαρκελόνης και της ευρύτερης περιοχής είναι μια θεμελιώδης και απαραίτητη υπηρεσία. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ε, ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούνται και τηρούνται πλήρως οι κανόνες ε, παροχής υπηρεσιών από τον ε, πάροχο. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών, να βελτιώσουμε τον έλεγχο της κατάστασης, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό μονοπόλιο. Από την άλλη, μάλλον δεδομένων όλων τούτων, πρέπει να μείνει ανοιχτή η αίτηση η αναφορά και να σταλεί στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για να λάβουν υπόψη τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ε, σε επίπεδο του δικαστικού του δικαστήριου στην Ισπανία. La verdad es que parece sensato, independientemente de la contradicción a la que ha llegado la justicia. Εκτός από αυτές τις αντιφάσεις ε, που προκύπτουν από το ισπανικό δικαστικό σύστημα, υπάρχει η στήριξη, ε, μάλλον τα δικαστήρια, ε, τα επιμέρους δικαστήρια στην Ισπανία έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Πρέπει λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά, προκειμένου να μπορέσουμε να την εξετάσουμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Να εξετάσουμε λοιπόν αυτές τις αντιφάσεις και να αποφασίσουμε τι μέλη Λέμε ότι το νερό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, είναι σαφές. Πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στο νερό. Ενδεχομένω να πρέπει να διασφαλίζεται από τον δημόσιο τομέα. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε εμείς αυτά τα ειχέγγυα ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κύριε Σαριάς. Eh, eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αρχίζω με ευχαριστίες προς τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ για την παρουσίαση. Άκουσα καταρχήν ότι αμφισβητείται η ισπανική δικαιοσύνη. Δεν επιτρέπεται να το δεχτώ αυτό, οπότε δεν συμφωνώ με την ουσία. Υπάρχει απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο εδώ, που είναι το ανώτατο όργανο της δικαστικής εξουσίας στην Ισπανία. Υπάρχει απόφαση. Δεν, είναι, δεν συνεχίζεται η διαδικασία, έχει κλείσει, υπάρχει απόφαση. Οπότε δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε απόφαση των του δικαστηρίου σε κράτος μέλος. Ε, είπαν ε, ότι χρειάζεται συζήτηση, ενώ υπάρχει απόφαση δεν υπάρχει απόφαση ακυρωτική. Τώρα για τις αποφάσεις. Να πω, παρακαλώ, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν οι αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση είναι από το, Ευρωπαϊκό Ανώτατο, από το Ανώτατο Ισπανικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό, Δικαστή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να ανατρέψει την απόφαση αυτή. Αυτό μπορεί να γίνει ενδεχομένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όχι όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αμφισβητήσει απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου μιας χώρας. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Επίσης το Κοινοβούλιο δεν έχει και την αρμοδιότητα να επανεξετάζει αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου. Και αν συνέβαινε αυτό θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας, το οποίο θα οδηγούσε σε χάος. Και συνεχώς θα ανατρέπονταν αποφάσεις. Όπως είπε ο κύριος Σαλίμπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να εξετάζουμε την αναφορά αυτή στο Κοινοβούλιο. Πρέπει σαφώς να κλείσει η αναφορά αφού ήδη υπάρχει απόφαση του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αν θέλουμε να το... Αν ε, θέλουν να το τραβήξουν περισσότερο, δεν πρέπει να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας πάνε στον ανάλογο φορέα. Ο κύριο Σουρτασούν. Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα που υποβλήθηκε στο ανώτατο δικαστήριο από μια ομάδα ε, Ισπανών πολιτών και πρέπει να αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, είναι ανοιχτή. Φανταστείτε, αν κλείσουμε την αναφορά αυτή τώρα και το ανώτατο δικαστήριο αποφασίσει να ακυρώσει τη δική του την απόφαση. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να κλείσουμε την αναφορά αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα να ακυρώσει το ανώτατο δικαστήριο την ίδια του την απόφαση. Νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον θα πρέπει να περιμένουμε για να επιληθεί το θέμα αυτό στην Ισπανία και μετά να πάρουμε απόφαση όντω. Ευχαριστώ κύριο Σάριας. Εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να κλείσει η αναφορά αυτή. Το λέει καθαρά η Κομισιόν στην απάντησή της ότι έχουμε μία ε, τελεσίδικη απόφαση. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο ε, βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής εναντίον της. Για να δώσουμε το λόγο στους ε, αναφέροντες για δύο λεπτά. Ευχαριστούμε τους ευρωβουλευτές που ήρθαν εδώ σήμερα για να πούνε τη γνώμη τους. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια πάνω σε αυτά. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η όλη αυτή η διαδικασία μας πάει πίσω στο 1953. Δόθηκε το συμβόλαιο αυτό ε, επί φραγκικού καθεστώτος. Ε, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ε, δεύτερον, μια άλλη εταιρεία παροχής ε, νερού ε, εταιρεία ίδρυυση, ζήτησε να αμφισβήτησε μάλλον αυτό το συμβόλαιο που ίσχυε από το 1953. Ε, εδώ ε, δεν υπάρχει θέμα τελεσίδικης απόφασης. Πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστηρίο πήρε μια απόφαση για τα ενυπόθηκα δάνεια η οποία τελικά ακυρώθηκε. Και πρέπει να σας πω ότι επί 8 χρόνια η εταιρεία αυτή έχει κόψει το νερό σε 75.000 οικογένειες. Πράγμα το οποίο ε, ε, υπονομεύει το ανθρώπινο δικαίωμά τους στο, στο νερό. Ευχαριστούμε. Εφόσον ακούσαμε την Κομισιόν, τους αναφέροντες και τα μέλη της Επιτροπής μας, η πρόταση είναι η εξής. Όπως είπαμε, υπήρξαν τέσσερις αποφάσεις από το Ανώτατο Δικαστήριο, όχι μία, τέσσερις αποφάσεις πήρε σχετικά το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν είναι ε, προς την Κομισιόν. Γνωρίζετε τίποτα γι' αυτό που αναφέρουν οι αναφέροντες σχετικά με την... Ε, ή μάλλον οι αναφέροντες γνωρίζουν ότι έχει υποβληθεί προσφυγή ακύρωσης ε, της ε, απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ε, ναι, διότι οι δικηγόροι μας της οργάνωσης που εκπροσωπούμε έχουν πει δημόσια ότι υπάρχει ε, δυνατότητα ακύρωση αυτή τη δικαστική απόφαση. Εμεί δεν ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αμφισβητήσει τι ε, εθνικέ δικαστικέ αποφάσει. Αυτό που ζητάμε από το Κοινοβούλιο είναι να εξετάσει αυτό το θέμα από την οπτική γωνία του ελεύθερου ανταγωνισμού, των κανόνων του ανταγωνισμού. Και άλλε επιχειρήσει ζητάνε το ίδιο. Πρόεδρο, να διευκρινίσω το εξή. Η Επιτροπή Αναφορών σέβεται πάντα τις τελικές αποφάσεις, τελεσίδικες αποφάσεις των κρατών μελών. Ε, σε αυτό το σημείο η Επιτροπή Περιφερειών πάντα κλείνει την αναφορά όταν υπάρχει τέτοια απόφαση του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου. Ε, επιπλέον, οι, μεγάλ, οι δύο μεγάλες εδώ πολιτικές ομάδες ΕΛΚ και σοσιαλιστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Η δική σας αναφορά σχετίζεται αποκλειστικά στην ίδρυυση της Βαρκελόνης και ε, ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει πάρει μια, ένα ισπανικό δικαστήριο, συγγνώμη, ε, έχει πάρει τη σχετική απόφαση. Ε, τώρα εσείς αναφέρεστε σε μια άλλη αναφορά που έχει να κάνει με, τον, με τις ανταγωνισμού. Αυτή θα πρέπει να, είναι μια, να υποβάλλετε μια άλλη αναφορά για αυτό το θέμα. Γιατί η αναφορά σας φαίνεται να ε, μιλάει για την ίδρυψη της Βαρκελόνης, ε, όπου δεν υπάρχει πλέον ε, περιθώριο αμφισβήτησης. Λοιπόν, η θέση μας ως Προεδρείου, λαμβάνοντας υπόψη την θέση της Κομισιόν και των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων, θα ήταν να κλείσουμε αυτή την αναφορά και προς τους αναφέροντες ε, θα έλεγα ότι μπορείτε να υποβάλλετε μια άλλη πιο γενική αναφορά σχετικά με την εκχώρηση συμβολέων ίδρευσης ε, ε, σε σχέση με τις συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτό όμως θα ήταν μια άλλη αναφορά. Γιατί υπάρχουν διάφορες αναφορές που έχουν υποβληθεί ε, για αυτό το θέμα. Αλλά ε, στη δικιά σας περίπτωση η αναφορά σας μιλάει για την ε, Σύμβαση Ίδρευσης της Βαρκελόνης. Για το θέμα αυτό υπάρχει ήδη τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Η Επιτροπή όμως αναφορών έχει την πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερι ειδικέ αποφάσει του Ανώτατου Δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Προτείνουμε να κλείσει λοιπόν η αναφορά. Έχω μία πρόταση, λέει ο κύριο ε, Ούρτασούν. Υπάρχει απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο επί αυτής της αναφοράς, αλλά υπάρχει και αίτημα κύρωσης τη απόφαση. Θα ήταν πιο σόφρον να δούμε τι θα γίνει και μπορούμε να συζητήσουμε σε επόμενη συνάντηση των συντονιστών και να το εξετάσουν το θέμα και οι πολιτικές ομάδες. Η δική μου πρόταση είναι αυτή. Γιατί μπορεί η αίτηση για ακύρωση να γίνει δεκτή από το ανώτατο δικαστήριο, ενώ εμείς θα έχουμε κλείσει πρόωρα την αναφορά. και θα μπορούμε να αποφασίσουμε. Εγώ προτείνω να περιμένουμε λίγο και να αποφασίσουμε σε μια συναδρίαση των συντονιστών. Αν αρνηθεί το ανώτατο δικαστήριο την ακύρωση, λύγει το θέμα. Μισό λεπτό κύριε Άριας. Κύριε Σαλίμπα, αν συμφωνείτε, είναι να δώσω με άλλον ένα μήνα στους αναφέροντες που είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη να τους δώσουμε ένα μήνα για να παρουσιάσουν την αίτηση ακύρωσης και να την παρουσιάσουμε στους συντονιστές. Η πρότασή μου σήμερα είναι να μην κλειστή αναφορά, αλλά να δώσουμε διορία ένα μήνα στους αναφέροντες να παρουσιάσουν την αίτηση ακύρωσης. Να πάρει το δρόμο της και να δούμε να Εμείς έχουμε τις πληροφορίες για τις ε, αποφάσεις. Αν δούμε ε, τι θα γίνει σε ένα μήνα, ε, θα αποφασίσουν οι συντονιστές. Ή θα κρατήσουν κλειστή ή θα ξανανοίξουν αυτή την αναφορά. Ο κύριος Αρίας. Αρίας, εντάξει. Ωραία. Έτσι θα κάνουμε. Οι αναφέροντες δεν είμαστε εμείς που υποβάλαμε το αίτημα κύρωσης. Θα δούμε αν η εταιρεία που το παρουσίασε μπορεί να μας δώσει την ενημέρωση ε, ή μπορεί να σας στείλουν απευθεία τις πληροφορίες. Δεν μπορούμε να στείλουμε επιστολή σε τρίτο μέρος που δεν είναι παρόν και δεν είναι και ενδιαφερόμενο μέρος στην υπόθεση γιατί θα παραβιάζαμε την προστασία των δεδομένων. Εγώ σας δίνω εσάς την ευκαιρία να κάνετε αυτό που πρότεινε ο κύριος Σουρτασούν και μετά θα αποφασίσουν οι συντονιστές. Η ε, διαδικασία της Επιτροπής Αναφορών πάντα έτσι ήταν από την αρχή, ότι όταν υπάρχει δηλαδή απόφαση από ανώτατο δικαστήριο μιας χώρας, κλείνουμε την αναφορά. Ευχαριστώ, λέει ο αναφέρον. Εμείς γνωρίζουμε από τα μέσα ενημέρωσης το αίτημα για ακύρωση. Δεν είχαμε άμεση ενημέρωση, αλλά θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Εγώ κλείνω τώρα την αναφορά και έχετε διορία ένα μήνα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την προσφυγή. Εγώ έχω τις τέσσερις αποφάσεις του του δικαστηρίου που υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να δει το φάκελο να τον ζητήσει. Ο κύριος Άριας, για να ξεκαθαρίσουμε τι συμφωνήσαμε. Η απόφαση τότε θα ληφθεί αυτομάτως, εάν πάρουμε την ε, τεκμηρίωση. Ναι, κλείνει η αναφορά. Αν πάρουμε την τεκμηρίωση μέσα σε ένα μήνα, μπορεί οι συντονιστές να ξανανοίξουν την αναφορά. Αυτό είναι δυνατόν στα πλαίσια των, των διαδικασιών μας. Κλείνει, σε ένα μήνα μπορεί να ξανανοίξουν την αναφορά οι συντονιστές. Νομίζω ότι είναι πολύ θεμητή αυτή η διαδικασία. Τελειώσαμε αυτό και προχωρούμε στο σημείο 21. α αλλαγή Όχι, το 22 θα πιάσουμε τώρα. Γιατί έχουμε μαζί μας τους Ιταλούς αναφέροντες, ενώ η αναφέροντα για το 21 δεν έχει έρθει. Λοιπόν, θα πάμε στο 22. Μικρόφωνο. Ε, και εμείς, για το, εμείς είμαστε εδώ επίσης και ήρθαμε για την 21. Το σημείο 21. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί ε, ευρωβουλευτές που θέλουν να προλάβουν. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι στην, ψηφίζουν στην Επιτροπή μκο. Γι' αυτό αλλάζουμε τη σειρά. Γι' αυτό είπαμε να αλλάξουμε τη σειρά. Okay. Ok, benvenuti. Adesso stiamo nel punto 22 che la petizione... Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο σημείο 22 στην αναφορά του 2017 0811 ε, εκ μέρους του Τζοβάνι Κορτέζε, Ιταλής ε, υπηκότητας, εκ μέρους της Ασοτζετσιόν Innovativo Δημοκράτικο, σχετικά με την κατασκευή δύο ε, λεκανών απορροής για το, στον ποταμό Σεβέζο. Ποιος είναι ο αναφέρον?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 Τούτο πώς Όλα εντάξει. Καλώς ήρθατε. Έχετε πέντε λεπτά για να παρουσιάσετε την αναφορά σας. Έχετε το λόγο. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Καλημέρα. Είμαι ο Τζοβάνι Κορτέζε και παρουσιάζω την αναφορά που συζητείτε για τις δεξαμενές αυτές. Ε, οι πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, είναι τρεις. Τεχνικό επίπεδο, επίπεδο που αφορά την υγιεινή και ε, τις παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Ε, και το τρίτο είναι ε, επίδραση στην υγεία των πολιτών. Για το, ένα, το σημείο 1 υπάρχουν διάφορα κρίσιμα και προβληματικά σημεία στον σχεδιασμό, ιδίως σχετικά με την γυτνίαση με το πάρκο Γκροάνε και το οικολογικό γενικά περιβάλλον, του, ε, της Λομβαρδίας, όπου ε, υπάρχει αυτό το πάρκο 17 εκταρίων. Επίσης, έχει να κάνει με τη λεκάνη απορροής που βρίσκεται πιο ψηλά από, το, από τη στάθμη των δεξο, δεξαμενών αυτών. Ε, υπάρχει ένα, μια έλλειψη του γεωλογικού φράγματος που προβλέπουν οι παραγωγοί και οι δεξαμενές αυτές επηρεάζουν και βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους καταναλωτές, σε σούπερ μάρκετ, στους πολίτες. Δεν εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των πολιτών. Σημείο 2. Ε, προβλήματα σχετικά με την ε, η, υγεία. Ε, ένας ε, καθηγητής το 2018 ε, μελέτησε το πόσο επηρεάζεται ο υδροφόρος ορίζοντας του Μιλάνου από την ε, κατασκευή του έργου αυτού και τι ε, αρρώστιες απειλούν τους πολίτες. Ε, υπάρχουν ε, καρκινογενέσεις, προβλήματα με το νοσοπικό σύστημα, στοιχεία καρκινογόνα, τετραχροθυλένιο, χλωρομεθάνιο, ε, και μια σειρά από άλλες ουσίες. Ε, πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες που είναι καρκινογόνοι, τετλαχρολοεθάνιο, νευροτοξικό. Ε, μετά, τα ύδατα του Σεβέζο, λόγω της ανάδευσης που γίνεται φέρνουν στην επιφάνεια αποθέσεις που υπάρχουν ως ειζήματα. Σημείο 3. Βιολογικά ε, προβλήματα. Τα βιολογικά προβλήματα ε, παρουσιάστηκαν από την κυρία Μαρίνα Κορτέζε, που είναι ειδική βιολόγος και που αναφέρεται σε τρεις μόνο από τις ουσίες που ε, είναι σχετικές. Το χλωρομεθάνιο, που είναι καρκινογόνο, είναι μια ουσία που βρίσκεται σε υγρή μορφή, σε ε, στα γλυκά ύδατα, χρησιμοποιείται σε, στη βιομηχανία βερνικιών, ε, επικάθεται νεφρούς. Γι' αυτό μπορεί ε, εξάλλου εύκολα να εισπνευθεί, ακόμα και για τα ζώα είναι επικίνδυνο. Ε, αναπτύσσονται ε, τοξικά αέρια όπως μονοξίδιο του άνθρακα και κιάνιο Εξάλλου, ε, πρόκειψε για μια ε, τροποποίηση της οδηγίας ε, που αφορά την κατασκευή και την παρασκευή και δημιουργή και εμπορία αυτού του αυτής της ουσίας. Μετά, υπάρχει ε, μια άλλη ουσία που ανήκει στην οικογένεια των χρονοτριαζινών, ε, μπαίνει μέσα στην διατροφική αλυσίδα, ε, διατηρείται στην, στο έδαφος για πολλά χρόνια και είναι διαταράκτης του ενδοκρινικού συστήμα, ενδοκρινολογικού συστήματος, προκαλεί λευχαιμία, μυελώματα, τρίτον, η γλυφοζάτο γλυφοζάτη. Ε, η ουσία αυτή κατατάσσεται με βάση την οδηγια 67548 67-548 ε, ως ε, επικίνδυνη για το περιβάλλον ε, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στα μάτια, ε, είναι τοξική για το περιβάλλον, για, το, ε, για τα ύδατα, χαρακτηρίζονται ως R51, R53, προκαλεί αύξηση της πίεσης, καρδιολογικά προβλήματα, επηρεάζει το χρωματόσωμα 430, ε, με αποτέλεσμα την ε, αποδόμηση των ιστών ε, και έχει δοθεί αποζημίωση 200 εκατομμύρια δολάρια για μια τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, από το 2018 προέκυψαν διάφορα γεγονότα. Το συμβόλαιο ε, αποφασίστηκε ε, μάλλον καταργήθηκε, ακυρώθηκε και ξεκίνησε νέος διαγωνισμός. Ε, επίσης, το 2019 ε, έχουμε νέες εξελίξεις αλλά το σχέδιο του διαγωνισμού αυτού είναι ίδιο με το προηγούμενο, αλλά χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Και υπάρχουν διάφορες επιτροπές νόσης πολιτών που εμπλέκονται στη διαδικασία τον Νοέμβριο του 2019 έγινε μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν 400 άτομα. Ε, οι θέσεις μας είναι αυτές του 2018. Δηλαδή να γίνει απορρίπανση των υδάτων του Σεβέζο σύμφωνα με το διάταγμα 152 του 2006 που αφορά την προστασία του ρήγματος ε, πριν γίνουν τα έργα, ό,τι διαφορετικά δεν θα είχε νόημα. Επιτρέψτε μου δύο ερωτήσεις. Η προστασία της υγείας είναι ή δεν είναι ένα ιερό και απαραβίαστο δικαίωμα των πολιτών και είναι ή δεν είναι καθήκον των ε, οργάνων των θεσμικών να προστατεύουν την υγεία των ε, πολιτών. Πρέπει να ε, ενεργήσουμε τώρα, να μην περιμένουμε για να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και αυτής της γενιάς αλλά και των επόμενων γενναίων. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή δουλειά. La la signora Laura Tabellini. Η κυρία Λάρα Ταμπελίνη από την Επιτροπή. Thank Ευχαριστώ. Καλημέρα. Το έργο στο οποίο αναφέρει ο αναφέρον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη ε, οδηγία EIA. Πράγματι, ε, αποτέλεσε αντικείμενο τη διαδικασία υπό αυτή την οδηγία. Και έτσι θέματα όπω ο αντίκτυπο τέτοιων έργων στην ανθρώπινη ζωή, στον εδροφόρο ορίζοντα, στην υγεία μάλλον, στο περιβάλλον και η εξέταση εναλλακτικών λύσεων φυσικά και θα πρέπει να εξεταστούν στη διαδικασία αυτή. Όμω, στην τελική επιλογή και στην τελική απόφαση για τα επιμέρου έργα και κατά πόσο θα πρέπει να αδειοδοτηθούν ή όχι, όλα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Να σημειώσουμε επίση ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο έργο, σε σχέση με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικέ αρχέ είναι σε θέση να ε, αξιολογήσουν την κατάσταση και να παρέμβουν αν αυτό είναι απαραίτητο. Η Επιτροπή επικεντρώνει τη δράση της σε ε, ζητήματα ευρύτερων πρακτικών ε, και συστηματικών στατιστικών στοιχείων και κατά πόσο συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο δεν ισχύει εδώ πέρα. Υπάρχει επάρκεια τη διαδικασία CIA σε αυτά τα ζητήματα και υπάρχει και έκθεση. Με βάση την οδηγία, εθνικέ αρχέ θα πρέπει να διασφαλίζουν τις, ε, την ποιότητα των εκθέσεων αυτών. Η οδηγία επίση αναφέρει συγκεκριμένη πρόσβαση ε, σε ένδικα μέσα, τα οποία θα πρέπει να είναι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο για την πλήρωση των σκοπών της οδηγίας. Με βάση των τις πληροφορίες που αναφέρονται, πράγματι υπήρχαν μια σειρά νομικών υποθέσεων στα εθνικά δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Κάποιες αφορούν την νομιμότητα των... της διαδικασίας υπό την οδηγία. Αυτές που πήγαν στο Τριμπουνάλιο Superiore ε, ε, καταρρίφθησαν και δεν υπάρχει ε, λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αμφισβητήσει τις ε, δικαστικές αποφάσεις της Ιταλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εγείρει ανησυχίε ότι έχει να κάνει με την κατάσταση ε, στον ποταμό Σφέρζο. Υπάρχει οδηγία περί ύδατος για αυτό το ζήτημα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια διαχείρισης των υδάτων και να συμπεριλαμβάνουν μέτρα, ούτω ώστε ε, να υπάρχει καλή ποιότητα του νερού σε όλο τον υδροφόρο ορίζοντα. Με προθεσμία το 2015. Όμω, σε ορισμένε περιπτώσει, τα κράτη-μέλη μπορούν να επεκτείνουν αυτό το χρονικό περιθώριο για την επίτευξη του στόχου. Βάσει των στοιχείων που έχουμε για την ευρύ... ε, με βάση το σχέδιο για την ποιότητα του νερού και του εδρυφόρου ορίζοντα ε, στην ευρύτερη περιοχή που συμπεριλαμβάνει και αυτό το ποταμό, ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν σχέδια για την επίτευξη αυτού του καλού επίπεδου μέχρι το 2027. Επομένως, δεν υπάρχουν ενδείξεις για, για την παραβίαση του, ε, της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. Τέλος, ο αναφέρον μιλάει και για την συμμόρφωση με, την, ε, με, άλλη οδηγία ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των αποβλήτων. Εδώ υπάρχουν τρεις διαδικασίες σε παραβάση κατά της Ιταλίας που μεταξύ άλλων έχουν να κάνουν και με την Λομβαρδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει τις απαραίτητε ενέργειε στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών επί παραβάση, προκειμένου οι παραβιάσεις αυτές ε, ως προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να σταματήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει ε, τις ενέργειές της για αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαλίβα. Ευχαριστώ. Σε αυτή την ε, περίπτωση δεν συμφωνώ με τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ποταμή είναι πολύ σημαντικό τμήμα του οικοσυστήματός μας και αφήνουν και πολύ σημαντικό αποτύπωμα στις κοινότητε μας. Ο ποταμός Σέβεσο επίσης είναι αναπόσπαστο τμήμα της ε, περιφέρειας Λομβαρδία. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να μην προβούμε σε ενέργειες, παρότι υπάρχει η αξιολόγηση αντικτύπου. Και από ό,τι έχουμε δει, πραγματικά δεν είμαι σίγουρος ότι όλα έχουν γίνει όπως πρέπει. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια λοιπόν και να αφήσουμε αυτές ε, τις κοινωνίες, τις τοπικές κοινωνίες μόνες τους. Γιατί υπάρχει πολύ σημαντική πίεση από αυτό το Δήμο, από τους πολίτες, διαμαρτύρονται κατά αυτών των έργων. Έχουμε τις πληροφορίες και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και θα υπάρξει μεγαλύτερο άχθος για τον ποταμό Σέβισο. Γι' αυτό όσους σοσιαλιστές και δημοκράτες θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία αυτού του πολύ σημαντικού ποταμού. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, πολύ σημαντικός φυσικός πόρος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε την περιφέρεια της Λομβαρδίας. Πρέπει λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να αποσταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Okay, thank you. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Συμφωνώ ε, να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, γιατί θα έχουμε μια δεύτερη ακρόαση των υπογραφώντων που θέτουν το πρόβλημα αυτό που πλήττει ιδιαίτερα τη βόρεια περιοχή του Μιλάνου εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένα έργο το οποίο προχώρησε, πρέπει να το πούμε και αυτό, με ελάχιστη προσοχή από τις ε, τοπικές αρχές και χωρίς να ακούσουν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εναλλακτικέ ε, λύσεις. Οι υπογράφοντας την αναφορά και άλλοι ε, αξιόπιστοι φορείς ή ενώσεις πολιτών έχουν υποβάλει τέτοιες εναλλακτικέ λύσεις και δεν εισακούστηκαν. Είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα από τις πλημμύρες του Σέβεζο στην περιοχή του Μιλάνου. Αλλά είναι μια ε, λύση, αυτή που, που επιλέχθηκε, που δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής και που θα ε, τσιμεντοποιήσει ακόμα περισσότερο ένα περιβάλλον ε, ήδη αρκετά επιβαρημένο, ενώ υπάρχουν λύσεις πολύ πιο αηφόρες και κατάλληλες. Ε, Παραδείγματος χάρη φυσικοί χώρη ε, περιορισμού των υδάτων όταν πλεονάζουν και ακριβώ όπω είπε και ο αναφέρον, εξυγίανση των υδάτων. Εμεί, σαν πρώτο στόχο, πριν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι τα ύδατα θα είναι καθαρά, ότι το νερό θα είναι καθαρό. Συμφωνώ και με τον συνάδελφο. Λυπάμαι που ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι όλα πάνε ε, καλά, όταν τα κράτη-μέλη επικαλούνται ε, διατάξεις που τους δίνουν ε, δυνατότητα παρέκκληση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων ε, από, από αποφάσεις που ελήφθησαν το 2015 και πάνε μέχρι το ε, μέλλον. Είναι πραγματικά λυπηρό να πρέπει να δεχτούμε θέσεις που πάνε τόσο μακριά στο χρόνο. Και όσον αφορά το ίδιο το έργο, θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το έργο, αυτές οι τεράστιες δεξαμενές που εξάλλου οι τοπικές αρχές ε, δεν ξέρουν να ε, πούνε καν αν θα είναι μία ή δύο, ε, ποιος ε, τις χρηματοδοτεί κλπ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μία από αυτές τις δεξαμενές θα κατασκευαστεί μέσα σε ένα πάρκο πράσινο 17 εκταρίων που αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον τόσο τσιμεντοποιημένο με τόσο πυκνό πληθυσμό που έχει τόσο μεγάλη ατμοσφαιρική επιβάρυνση γιατί η λεκάνη της Πανανίας ε, ε, έχει ε, ατμοσφαιρικές συνθήκες που είναι χειρότερες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ευρώπης. Και έχουμε μια οδηγία σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και αυτό ε, εξίζει να ληφθεί υπόψη. Είναι κάτι το παράλογο, κάτι που δεν έχει νόημα η επιλογή αυτού του έργου. Ο κίνδυνος ε, ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα ύδατα ε, ε, του Σεβέζο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο, διότι διαφορετικά ε, τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Με όλες αυτές τις επικίνδυνες και τοξικές ουσίες για τις οποίες μας μίλησε ήδη ο αναφέρον. Επαναλαμβάνω επίσης ότι αυτό που έχει λείψει από αυτό το έργο, αυτό που λείπει είναι μια ε, ένας πραγματικός και ανοιχτός ε, και συμμετοχικός διάλογος με τους πολίτες. Ε, οι αρχές ήταν κλειστές, κοφεύουν απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή. Έχουμε στείλει επιστολές ε, σε τοπικές και περιφερειακές αρχές και στην περιφέρεια της Λομβαρδίας και στην πόλη του Μιλάνου. Η περιφέρεια της Λομβαρδίας ε, έστειλε μια απίστευτη πραγματικά απάντηση ε, λέγοντας περίπου not in my backyard, ε, αυτό ήταν το νόημα α, α, της απάντησης, δηλαδή αυτό ε, υποτίθεται ότι ενοχλεί ε, τους αναφέροντες, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι δεν θέλουν στη γειτονιά τους ένα τέτοιο έργο, είναι ότι ε, θέλουν να προστατευτεί η υγεία και, και το περιβάλλον μιας περιοχής που είναι πάρα πολύ επιβαρημένη, όπως είπαμε. Ε, οι αρχές τη του, της πόλης του Μιλάνου δεν απάντησαν ποτέ. ζητάω λοιπόν και εγώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να ε, επαναλάβουμε αποστολή ε, τέτοιων επιστολών ε, και στο Δήμο του Μιλάνου και στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Και θεωρώ, τώρα που έχουμε τη νέα επιτροπή της ε, κυρίας Βαντερ Λάιεν, ε, ε, θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και στα θέματα του κλίματος και αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη με προστασία όλων αυτών των περιοχών της Ευρώπης που κινδυνεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο Αναφένο για δύο λεπτά. Εμείς ε, θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει εδώ πέρα από τις μεγάλες αυτές τρύπες που ανοίγονται. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, το έδαφος, το περιβάλλον και οι πολίτες με την δέουσα προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές λύσεις έχουν όμως εδώ επικεντρωθεί μόνο στην κατασκευή αυτών των δεξαμενών και τίποτα άλλο. Με τις τεράστιες αυτές εξκαφές εκατομμυρίων ε, κυβικών μέτρων ε, ε, χώματος που μετακινούνται. Γιατί αν γίνουν αυτές ε, οι δεξαμενέ για την υγεία των πολιτών μας, των παιδιών μας, των εγγονιών μας, τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Γι' αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο να κάνουμε κάτι και σας το έγραψα εξάλλου. Δεν είναι δυνατόν να ε, συζητείτε το θέμα αυτό χωρίς να λαμβάνετε υπόψη ε, η Υγεία των Πολιτών, η ίδια η ΆΙΠΟ της Λομβαρδίας ε, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρονται αυτοί για την ε, Υγεία των Πολιτών. Απλώς αντιμετωπίζουν το έργο αυτό ως ένα υδρολογικό έργο. Δηλαδή, πολίτες δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Ε, δεν έχουν λόγο. Είτε, είτε το θέλουν είτε όχι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σας ζητάμε βοήθεια για την υγεία των ε, ε, πολιτών. Εντάξει, μπορείτε να πείτε ότι εγώ τα έχω τα χρονάκια μου, αλλά ε, σκεφτείτε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τον αναφέροντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής. Η πρότασή μας είναι να μην ανοιχτεί η αναφορά, να αποσταλεί, να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Περιβαλλοντικών Υποθέσεων για περαιτέρω πληροφορίες και να υπάρξει μια επιστολή προς τις περιφερειακές αρχές στη Λομβαρδία και το Λιμιλάνο, ε, και να του ενημερώσουμε για τι πληροφορίε που μας παρέχει ο αναφέρον και τι εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να ζητήσουμε διευκρινήσει για τα επόμενα μέτρα που θα υιοθετηθούν σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αναφέροντα. Λοιπόν, επι, επανερχόμαστε στο σημείο 21 το οποίο προσπεράσαμε προηγουμένως. 865 κάθετος 18 ε, της κυρίας Βαγιουνοτόβα εξ ονόματος ε, του Κέντρου Ανεξάρτητης Διαβίωσης για την χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Βουλγαρία. Είναι εδώ οι αναφέροντες. Καλώς ήρθατε. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για να κάνετε την παρουσίασή σας και μετά θα σας ξαναδώσουμε στο τέλος του γύρου τραπέζι σε άλλα δύο λεπτά. Θα μιλήσει ένας ή δύο. Εντάξει, δυόμιση λεπτά λοιπόν ο καθένας. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ονομάζομαι Ανέτα Γιάννοβα Ελσόμβα και αντικαθιστώ εδώ την ε, Κάπκα Παναγιώτοβα που δεν ε, μπορούσε να ε, παραβρεθεί εδώ σήμερα. Ήθελα να σας μιλήσω για το τι συμβαίνει στον χώρο των ατόμων με αναπηρία στη Βουλγαρία το 2005. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Η βουλγαρική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την κατασκευή ε, κτηρίων και οικοδομημάτων για παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες και για ηλικιωμένους. Παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης. Στη Βουλγαρία αυτό σημαίνει ότι αντικαθιστώνται έτσι τα παλαιότερα μεγάλα ιδρύματα με μικρότερα ε, μικρότερους οίκου ευγυρία ή ε, άλλες δομές ε, φροντίδας ε, των ατόμων με αναπηρία και το καθεξής. Εκατοντάδες τέτοιες έχουν οικοδομηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Στι νέε αυτές δομές έχουμε την ίδια νοοτροπία που γνωρίζουμε από τα μεγάλα ιδρύματα, που απλώς μεταφέρεται σε μικρότερες δομές. Έχουμε νέα οικοδομήματα λοιπόν, μικρότερο μέγεθος των εγκαταστάσεων και ε, μικρότερο αριθμό ατόμων που διαμένουν εκεί, αλλά τίποτα άλλο δεν αλλάζει. Μετά από 10 χρόνια επενδύσεων βλέπουμε ότι η αποϊδρυματοποίηση για τα παιδιά στη Βουλγαρία φαίνεται επιτυχής μόνο για όσου δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά ακόμα βρίσκονται απομονωμένα, στερούνται των θεμελιωδών του δικαιωμάτων, πλήττονται από αυτό το ιδρυματικό μοντέλο και χωρίς ε, την, χωρίς την απαραίτητη αποκατάσταση από το τραύμα το οποίο έχουν υποστεί. Η διαδικασία της ε, αποδηματοποίησης αφορά τα κτίρια και όχι τους ανθρώπους. Έχουμε εδώ ένα σύντομο βίντεο. Um, there is some sound there. Κανονικά έχει και ήχο. Uh, this picture are... Όμως ε, και οι εικόνες ε, μιλούν από μόνες τους. Είναι ένα βίντεο το οποίο φτιάξαμε πέρυσι τον Οκτώβριο. I, I took part in this uh, uh, visit Κατά τη διάρκεια μια επίσκεψη σε διάφορα ιδρύματα στην Βουλγαρία, συμμετείχα και εγώ προσωπικά και τα είδα όλα οι And I have say that there is a lot of uh, torture and... Και μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά αυτά βασανίζονται, παραμελούνται. Όλα αυτά τα εκτήρια είναι πολύ όμορφα απ' έξω, αλλά στην ουσία είναι αποτροπιαστικά. We have another side. Okay. After 10... Μετά από 10 χρόνια επενδύσεων λοιπόν σε τέτοιες ε, ομαδικές ε, δομές για παιδιά και νέους, η κυβέρνηση τώρα προετοιμάζεται να κάνει ακόμα περισσότερες δαπάνες για το ίδιο μοντέλο ή ακόμα και χειρότερο για τους ενήλικες. Σχεδιάζει λοιπόν η κυβέρνηση να ε, κατασκευάσει 68 τέτοιε ομαδικέ οικίε και θα επηρεάσει τουλάχιστον 1.020 άτομα χωρί καμία ε, διασφάλιση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Είναι σαφέ ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί απλώ θα μεταφερθούν από το ένα ίδρυμα στο άλλο και όλο αυτό υποστηρίζεται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να συνεχίσω και εγώ να σας παρουσιάσω το νομικό υπόβαθρο. Κανονικά λοιπόν επί χάρτου προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε να κάνουμε εδώ με την ε, ε, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε, πιο συγκεκριμένα το άρθρο 19, και υπάρχουν γενικέ παρατηρήσει που πρόκειται για ερμηνείε ε, των ε, μεμονωμένων ανθρωπινών δικαιωμάτων που επεξηγούν τη σύμβαση. Μετά έχουμε την Σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρα 26-24, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για την Αναπηρία από το 2010 έως το 2020, ε, μια σειρά νομικών πράξεων που προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Να σα δείξω αυτή την γενική παρατήρηση 5 που μιλάει για μεγάλε ή μικρέ τέτοιε ομαδικέ κατοικίε που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνε για παιδιά γιατί δεν υπάρχει υποκατάστατο για αυτά τα παιδιά σε σχέση με την ανατροφή του στο πλαίσιο μια οικογένεια. Αυτά τα ιδρύματα λοιπόν δεν μπορούν να αποκαταστήσουν ε, μια οικογένεια. Έχουμε λοιπόν προτάσεις και συστάσεις αντί να δημιουργούμε νέα ιδρύματα και να παραβιάζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των ατόμων είναι σημαντικό να έχουμε εναλλακτικέ ε, λύσεις, να επενδύσουμε σε αυτές τις λύσεις, να στηρίζουμε ε, την διαβίωση αυτών των ατόμων μέσα σε μια κοινότητα. θα πρέπει να ε, επενδύσουμε και την πρόσβαση σε αυτά τα άτομα ε, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες. Έχουμε και ένα σύντομο βίντεο, αν μου επιτρέπετε, τριών λεπτών. Θα θέλαμε να σας το δείξουμε. Μπορούμε. If there is a sound. Αν μπορούμε να βάλουμε και τον ήχο. If there is a sound, it would be good. Εκτός μικροφώνου η πρόεδρος. What do we do then? We don't do mm. No. No, then, then okay, then no. We, yeah.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 I'm going to give Η Κομισιόν. Κυρία Λαγκρή Μπομών, ευχαριστώ για όλη αυτή την παρουσίαση και την προσφορά προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία. Έχει γίνει συζήτηση και πολλές ανταλλαγές ήδη. υπάρχουν κάποια συμπεράσματα και θα δώσω και ορισμένα παραδείγματα πρόσθετα στοιχεία που δεν, που δεν σημαίνουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και πρέπει κατεπηγόντως σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβουμε δράση. Στη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει υποστήριξη ε, στους ανθρώπους αυτούς ώστε να ζουν ανεξάρτητα και να διαβιώνουν μέσα στις κοινότητες. Υπάρχουν και 43 εκατομμύρια για τις υποδομές. Για πάνω από 150 εκατομμύρια δόθηκαν σε αυτή την περίοδο να πω ότι οι προσπάθειες δεν γίνονται μόνο ε, για τα κτίρια. Έχουμε 8.000 παιδιά σε ιδρύματα και περίπου 5.000 που μπήκαν σε οικογένειες ή σε συγγενείς. Πάνω από 2.000 παιδιά είναι σε ανάδοχες οικογένειες και αν τα στοιχεία μου είναι σωστά Υπάρχουν και 2.200-2.500 παιδιά σε φροντίδα οικογενειακή και 600 παιδιά μεταξύ αυτών είναι με αναπηρίες. 149 μικρά σπίτια, μικρές ομάδες όπως τα λέμε. Από τα 14 εκατομμύρια ε, έχουμε χρηματοδότηση σε ανάδοχη φροντίδα χρηματοδοτούν πολλά προληπτικά μέτρα για να προλάβουν τον ιδρυματισμό. Παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, κατάρτιση. Έχουμε επίσης και λειτουργίες στήριξης των νέων ε, ενηλίκων που φεύγουν από τα ιδρύματα για να τους βοηθήσουμε να χτίσουν το μέλλον τους ε, τους βοηθούν και οι ομολογοί τους. Υπάρχουν λοιπόν κονδυλία για να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία, προσπαθώντας να στηρίξουμε όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχουν και πολλές εναλλακτικέ. Δεν λέω ότι το οικογενειακό περιβάλλον για αυτά τα παιδιά δεν είναι βελτίωση, αλλά και ε, τα κονδύλια που είναι περίπου 150 εκατομμύρια είναι για αυτό που λέμε πατρονάς φροντίδα, για προσωπική βοήθεια, με προσωπικό δηλαδή βοηθό. Υπάρχουν πολλές ε, προσπάθειες και γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες αν δείτε όλο τον φάκελο 43 εκατομμύρια για τις υποδομές και την αποκατάσταση και ένα παρόμοιο ποσό για εναλλακτικέ λύσεις. Θέλω να διαφοροποιήσω λίγο αυτά που είδαμε, που ήταν βεβαίως πολύ συγκινητικές και ε, εντυπωσιακέ εικόνες. Θέλω να προσθέσω δύο ακόμα στοιχεία. Έγινε μία αξιολόγηση της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, γιατί τότε χρηματοδοτηθήκαν αυτά τα σπίτια που είδαμε και λένε ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις συμβάλλει πολύ στην ποιότητα ζωής των νέων που βοηθούνται με δραστηριότητες, ε, βασική ιατροφαρμακευτική φροντίδα, πρόσβαση σε διοικητικές διαδικασίες, που υπογραμμίζουν την ποιοτική αλλαγή για αυτά τα παιδιά. Βέβαια λέγουν ότι υπάρχουν ε, βελτιώσεις και έχουν και συστάσεις σε σχέση με τις ανάγκες εξατομικευμένης φροντίδας, πολύ παραγοντική προσέγγιση, ποιότητα και βέβαια και άλλα θέματα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά η εικόνα δεν είναι τόσο αρνητική από την άλλη πλευρά. Και προσωπικά πρέπει να πω ότι επισκέφτηκα δύο κέντρα οικογένειας, οικογενειακά. Οι πέντε έχουν ε, επισκεφθεί άλλοι συνάδελφοι, συνολικά έχουμε δει επτά και προσωπικά ε, εντυπωσιάστηκα από αυτά τα σπίτια που έχουν μια οικογενειακή δομή και μπορούν να συζητούν τα παιδιά, να συμμετέχουν στην κοινότητα. Λένε ότι στο πρώτο στάδιο ήταν πιο περίπλοκα τα πράγματα για να ανοίξει προς αυτές τις δομές η κοινότητα, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να βρίσκουν δραστηριότητες και να έχουν επαφές τα παιδιά με την κοινότητα και ειλικρινά πρέπει να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό, ήταν ένα διαδραστικό περιβάλλον. Μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό και αυτή η εικόνα, αλλά πάντως και εμείς προσπαθήσαμε να δούμε ε, από κοντά την κατάσταση και είδαμε ότι ασχολούνται πάρα πολύ, είναι δηλαδή αφιερώνεται το προσωπικό σε αυτά τα παιδιά, τα οποία υποστηρίζονται και ζουν ε, ευχαριστημένα μαζί. Πριν να σας δώσω το λόγο, θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό δεν το είδα στην αναφορά. Στα κέντρα υπάρχουν παιδιά τα οποία όμως τα φροντίζουν. Ποιος τα φροντίζει, οι γονείς ή το κράτος. Τα παιδιά σε αυτά τα κέντρα είναι παιδιά που δεν τα φροντίζει πια η οικογένειά, του, η οικογένειά τους. Ε, αν μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό, ίσως η Κομισιόν. Υπάρχουν πιο έμπειροι βέβαια εδώ για να απαντήσουν ε, οι, οι αρχές. Δεν μπόρεσαν εναλλακτικές για να πάνε τα παιδιά πίσω στις οικογένειες ή σε συγγενείς και λόγω της κατάστασής τους ε, δεν μπορούσαν να βρουν ανάδοχους γονείς. Δηλαδή ε, είναι παιδιά τα οποία είναι σε ιδρύματα. Το κράτος τα φροντίζει. Δεν τα φροντίζουν οι οικογένειες, δεν ε, έχουν αυτή την ευθύνη και οι αναφέροντες ζητούν όσο γίνεται περισσότερη υποστήριξη, βοήθεια για να πάνε ας πούμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Ωραία. Ήθελα απλώς να το ξεκαθαρίσω αυτό στο μυαλό μου. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά στο σύστημα αυτό καλύπτονται από το κράτος. Αλλά αν συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα σύστημα που ε, απομονώνει τα παιδιά, στο τέλος οι οικογένειες θα προσφεύγουν σε αυτήν την λύση. Και μετά θα είναι πιο δύσκολο οι οικογένειες να στηρίξουν σε οικογενειακό περιβάλλον το παιδί. Αυτό λέμε, αντί να επενδύσουμε σε ένα σύστημα όπως το παλιό που απομονώνει τα παιδιά, μπορούμε να επενδύσουμε σε συστήματα που δεν τα απομονώνουν και δεν τα αποκλίνουν. Και αυτό όχι επειδή τα παιδιά δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν υπάρχουν υποστηρικτικές δομές. Τα περισσότερα παιδιά έχουν οικογένειες και οι οικογένειες αυτές είναι πολύ φτωχές. Οπότε δεν ε, υποστηρίζονται πολύ φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να παρέχουν ε, φροντίδα στα παιδιά τους. Η ανάδοχη φροντίδα για παιδιά με αναπηρία σχεδόν δεν υφίσταται στην ε, Βουλγαρία. Και υπάρχουν κάποιες ανάδοχες οικογένειες που θέλουν να παρατείνουν ε, την ε, φροντίδα, αλλά λόγω προβλημάτων στην κοινότητα δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στη φροντίδα. Ο κύριος Αλίμπα. Ε, είναι πρόβλημα η έλλειψη οικογένειας, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την πραγματικότητα ε, και πώς ε, αυτή επιδρά στους πιο ευάλωτους. Πρέπει να τους εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα ζωής. Αν δεν το κάνουμε εμείς, αν δεν το αναλάβουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Καταλαβαίνω βέβαια τις δυσκολίες των κρατών μελών όπως η Βουλγαρία. Πρέπει να υπάρχει μία μετάβαση από ένα σύστημα ιδρυματοποίησης σε ένα σύστημα κοινοτική φροντίδας, που είναι και η καλύτερη φροντίδα και η καλύτερη βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως πιστεύω ότι χρειάζεται καλύτερη στρατηγική, πιο ισχυρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα απευθύνεται σε ανθρώπους με αναπηρίες. Πρέπει να έχουμε πιο μεγάλες φιλοδοξίες εδώ. Οπότε, όποτε ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών σε ένα κράτος μέλος, ε, κονδύλια που πάνε για άτομα με αναπηρία πρέπει να φροντίζουμε να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε μία μετατόπιση α, της φροντίδας από το Ίδρυμα στην κοινότητα. Δεν αρκεί αυτό, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και αυτά θα πρέπει να δίδονται για την βέλτιστη φροντίδα. Βλέπουμε όμως αυτά τα βίντεο στα νέα αυτά ιδρύματα που θα έπρεπε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να αποκτήσουμε ένα καλύτερο και σαφέστερο σχέδιο και να υπάρχει περισσότερη παρακολούθηση και έλεγχος, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές αναφορές που αφορούν άτομα με αναπηρία και νομίζω ότι προέρχονται περισσότερο από ορισμένα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες είδαμε πολλές αναφορές από τη Βουλγαρία που αφορούν ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καλύτερη στρατηγική από την πλευρά της Κομισιόν ώστε αυτά τα ευάλωτα πρόσωπα να έχουν καλή ποιότητα ζωής, την καλύτερη δυνατή που δεν παρέχεται αυτή τη στιγμή σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και τους αναφερόντες που έφεραν εδώ αυτό το ζήτημα και αυτές τις μαρτυρίες που μόλις ακούσαμε και είδαμε. Είναι πάντα βέβαια δύσκολο να ελέγξει κανείς τα συναισθήματά του μπροστά σε μια τέτοια θεσμική βία ε, στην οποία υποβάλλονται οι πιο ευάλωτοι από εμάς. Τα θεσμικά ιδρύματα ουσιαστικά στερούν από αυτά τα άτομα τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους. Κανείς δε μετά δεν είναι αυτόνομος, ε, τις επιλογέ που κάνουν στη ζωή του βρίσκονται απομονωμένοι, ιδρυματοποιημένοι και όλα αυτά με την έγκριση και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Το 2019 η Καταλήνα Βεντάρνες Γκουιά είχε, είχε ζητήσει το σταδιακό κλείσιμο όλων αυτών των ε, Ιδρυμάτων. Είναι λοιπόν απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξάνει τον αριθμό αυτών των ατόμων παρά τι ε, διεθνείς τη δεσμεύσει και τη Ευρωπαϊκή Χάρτα των Μελλονών Δικαιωμάτων. Η διαδικασία ε, μετάβασης από την ε, θεσμική φροντίδα σε μία ανάδοχη φροντίδα είναι περιπλοκή, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. στη Βουλγαρία εδώ και χρόνια η διαδικασία ε, είχε να κάνει με, την, ε, ε, με το κλείσιμο αυτών των ιδρυμάτων και την δημιουργία μικρότερων δομών. Όπως αναφέρεται όμως, βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει, ε, δεν έχει δοθεί τέλος στην απομόνωση αυτών των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων στη βουλγαρική κοινωνία. Όταν κάποιος δεν μπορεί να επιλέξει πού, με ποιον και με ποιον τρόπο θα ζει και όταν απλώς μεταφέρεται από ένα μεγάλο ίδρυμα σε ένα μικρότερο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποϊδρυματοποίηση. Πρόκειται απλώς για μια συνέχεια μιας πολιτικής απομόνωσης και παραβίασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Σήμερα μιλούμε για τη Βουλγαρία, αλλά να γνωρίζετε ότι αυτή η πρακτική υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη. Τα ευρωπαϊκά ταμεία χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο για την κατασκευή τέτοιων ιδρυμάτων μικρού μεγέθους όπως λένε. Αυτό συμβαίνει και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, στην Εστονία, στην Πορτογαλία, στην Πολωνία, στην Αυστρία και αλλού. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να δώσουμε ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να σεβαστούμε τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. θα ήθελα να πω ότι αυτή ε, η τοποθέτηση έχει να κάνει περισσότερο με το, με το κοινωνικό πλαίσιο. Το 63% των ατόμων με αναπηρία στην Γαλλία ε, μπαίνουν κανονικά στο σχολείο. Σε σχέση με το 42% ε, των νέων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Επομένω, η κοινωνική πολιτική έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ιδρυματοποίηση για ό,τι φορά τη διασφάλιση της ε, ισότητας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ε, ευκαιρίε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λάγκεν είπε «Ναι, ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να πάρω το λόγο. Δεν είμαι μέλο αυτή τη επιτροπή. συμμετέχω περισσότερο στην Επιτροπή απασχόληση. Λοιπόν, άτομα με αναπηρίε. Η ανεξάρτητη διαβίωση είναι μία απόδειξη των, ε, και δείχνει την ε, πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση. Έχει να κάνει με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιτρέπουν ε, στα άτομα με αναπηρία να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα Ιδρύματα δεν θεωρούνται υπηρεσίες με βάση την κοινότητα και δεν βοηθούν αυτά τα άτομα να διεξάγουν μια ανεξάρτητη ζωή. Κανένα Ίδρυμα δεν είναι καλό. Στο σημείο 5 της ε, σύμβασης στο ΙΕ, λοιπόν, αναφέρεται ότι ούτε τα μεγάλα ιδρύματα με πάνω από 100 άτομα, είτε τα μικρότερα με 5 με 8 άτομα, είτε τα μεμονωμένα, μεμονωμένες κατοικίες μπορούν να θεωρηθούν ε, διευθετήσεις ανεξάρτητες διαβίωσης αν υπάρχουν άλλα ε, καθοριστικά στοιχεία ιδρυματοποίησης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό βρίσκουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μεταφορά των τροφίμων, αν θέλετε, από τα μεγάλα στα μικρά ιδρύματα δεν είναι ανεξάρτητη διαβίωση ούτε από ιδρυματοποίηση. Απλώς του μεταφέρουμε το ένα ίδρυμα στο άλλο. Και έτσι συνεχίζουμε την παραβίαση και ευρωπαϊκού δικαίου και των εθνικού δικαίου δεν πρόκειται ούτε για μεταβατική κατάσταση. Ε, στοιχεία δείχνουν ότι πολλά παιδιά που μεταφέρονται σε μικρότερες δομές δεν φεύγουν ποτέ από αυτές. Η αποϊδραματοποίηση είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένως, γιατί πολλές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό μας λένε τα τελευταία 20 χρόνια. Ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά ταμεία και κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούνται για την ε, απομόνωση και, τον, ε, ε, και τις διακρίσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται και λοιπόν μια, για μια κακή πρακτική, δεν πρέπει να συμβαίνει πουθενά. Αυτό που γίνεται τώρα στη Βουλγαρία πρέπει να αναλάβουμε δράση και δεν πρόκειται για τεχνικό διαδικαστικό ζήτημα για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μιλούμε για ανθρώπινες ζωές και την παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χώσα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν είναι εύκολο να εξετάσουμε αυτή την αναφορά και, και να είμαστε ουδέτεροι. Είδαμε το βίντεο. Γνωρίζω την οργάνωση που υποβάλλει την αναφορά. Εδώ και χρόνια είμαστε σε επαφή και προσπίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα να σας καλέσω να είμαστε συνετοί. Ας μην ξεχνούμε ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ε, υπολείπεται σημαντικά των υπολείπων ε, ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι έχει να κάνει με την αποϊδρυματοποίηση και την ε, δημιουργία νέων συστημάτων φροντίδας που βασίζονται στην κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο παίρνει πολλή ενέργεια, πολλά χρήματα και προσωπική προσπάθεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι οι βουλγαρικές αρχές κάτι προσπαθούν να κάνουν. Έχω διαβάσει με μεγάλη προσοχή το υλικό που λάβαμε ε, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα και την παρουσίαση. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να υπήρχε η απαραίτητη βούληση, απλώς να μην επετέφθη ο τελικός στοχός, σκοπός. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ βουλγαρικών αρχών και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε και να εμπλέξουμε αυτές τις οργανώσεις στη διαδικασία αυτή και έχουμε δει ότι οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν συζητήσει τα θέματα σε αρκετό βάθος με τέτοιες οργανώσεις που προσωπούν άτομα με αναπηρία και ως εκ τούτου τα βήματα που έγιναν δεν ήταν τα απαραίτητα ε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία. Και πρέπει να διαρευνήσουμε αν αυτά τα βήματα συνάδουν και με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Το 2012 Εγώ ασχολήθηκα και μελέτησα σε βάθος το θέμα ε, των ευρωπαϊκών ταμείων σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία. Τώρα πλέον έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία και αυστηρού κανόνε. Τα κράτη-μέλη όμω έχουν ακόμα ένα περιθώριο ευελιξία και αυτό είναι το βασικό μέλημα μας εδώ. Το κράτος μέλος, οι κοινότητες αυτές και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό σύστημα φροντίδας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά και θα ήθελα να υπάρξει μια επιστολή ή ένα έγγραφο των βουλγαρικών αρχών. Θα ήθελα να ακούσουμε και την πλευρά των βουλγαρικών αρχών για αυτό το ζήτημα. Και αφού λάβουμε τέτοιες πληροφορίες, να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσει στι βουλγαρικέ αρχέ ή στι αρχέ των κρατών μελών να αξιοποιούν σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί αυτή τη στιγμή, με κάθε ειλικρίνεια, δεν μπορώ να πω αν οι βουλγαρικέ αρχέ χρησιμοποίησαν σωστά ή λάθο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ζητώ λοιπόν να ακούσουμε πρώτα και να ζητήσουμε τη θέση των βουλγαρικών αρχών και όταν λάβουμε αυτές τις απαραίτητε πληροφορίες και λεπτομερή επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νέα στοιχεία από τους αναφέροντες, να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούσουμε πρώτα πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές για να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις. Πρέπει να, το, να εξετάσουμε πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κάνεφ. Είναι και προσωπικό για μένα το θέμα και συναισθηματικά φορτισμένο γιατί εδώ και αρκετές δεκαετίες εργάζομαι με παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Ε, τη δεκαετία του 90 ε, είχα ασχοληθεί ως θελοντής και εξειδικεύτηκα στην προσπάθεια ένταξης στην κοινωνία παιδιών με σοβαρές αναπηρίες. Είμαι, γνωρίζω και είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι ο αντίκτυπος της ε, αποκλειστικής φροντίδας σε ένα παιδί με βαριά αναπηρία είναι τεράστιος. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μεγάλη πρόοδο. Τα παιδιά που είδαμε στο βίντεο δεν είναι καταδικασμένα να ζουν έτσι. Βεβαίως έχουν μια σοβαρή αναπηρία, αλλά μπορούν να προχωρήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι είδαμε. Και είμαι πεπισμένος ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, χρειάζεται ένας σε βάθος έλεγχος στα ολοκληρωμένα και συνεχιζόμενα έργα αυτού του τύπου στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Και πιο σημαντικό, χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση του ίδιου του μοντέλου ολόκληρου του μοντέλου. Στη δεκαετία του 90, όταν δουλεύαμε με τα παιδιά στα Ιδρύματα, ε, ήταν αυτά τα τεράστια κομμουνιστικού τύπου Ιδρύματα, απομονωμένα κάπου στην εξοχή. Και τώρα βλέπω και είμαι αντιπρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής του Εθνικού Κοινοβουλίου επίσης ήμουν και ξέρω πως ε, εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το ίδιο μοντέλο, μόνο που τα σπίτια, τα, οι κατοικίε είναι λίγο μικρότερες και σε καλύτερη κατάσταση, αλλά το μοντέλο δεν διαφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι αν δαπανώνται ε, ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για αυτή την ψεύδο αποκατάσταση και ολοκλήρωση, ε, δεν θα έχουμε αποτελέσματα θα έχουμε αποτελέσματα και στη Βουλγαρία και στις άλλες χώρες σαν αυτά που είδαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά, λέει ο κύριος Βιτανόφ. Σχεδόν τίποτα δεν έχω να προσθέσω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ήδη. Ε, συνυπογράφω και προσυπογράφω. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια πρόοδος έχει γίνει. Για κάποιον, ως κάποιος που ξέρει την κατάσταση επιτόπου θα ήθελα να πω ότι παρά τα σημαντικά κονδύλια που έχουν δοθεί δεν υπήρξε πραγματική αποϊδρυματοποίηση στη Βουλγαρία, τουλάχιστον όχι αυτού του τύπου που κατανοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπήρχαν τεράστια ιδρύματα πολύ μεγάλα. Έκλεισαν αυτά. Αλλά δεν άλλαξε τίποτε στο ίδιο το σύστημα, εις ό,τι αφορά δηλαδή την κοινωνική ένταξη. Απλώς πήγανε από μεγαλύτερα ιδρύματα σε μικρότερα ιδρύματα. Συμφωνώ απόλυτα με τους αναφέροντες. Πράγματι, άλλαξαν οι συνθήκες διαβίωσης, αλλά η ποιότητα ζωής παρέμεινε αμετάβλητη. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά είναι τεκμηριωμένη και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει πολλά να κάνει για να βοηθήσει ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γίνεται να σας δώσω για τα γρήγορα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είδαμε, ε, αυτή είναι μία μετάβαση που και γίνονται επενδύσεις σε μικρότερα ιδρύματα. Αλλά αυτό δεν είναι πραγματική μετάβαση. Η μετάβαση έγινε πριν από 20-30 χρόνια. Το να βάλεις από μεγαλύτερα σε μικρότερα ιδρύματα τους ανθρώπους αυτούς ε, συνιστά καταστρατήγηση των ε, ευρωπαϊκών προτύπων. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται μόνο στη Βουλγαρία, γίνεται και σε άλλες χώρες μέλη όχι μόνο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη Δυτική. Η Βουλγαρία ε, δείχνει την κατάσταση. Τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προστατεύονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Υπάρχει και μία υπόθεση τώρα που τρέχει στα δικαστήρια και θα δούμε τι απόφαση θα βγει. Λοιπόν, ακούσαμε τους αναφέροντες την Κομισιόν και μέλη της Επιτροπής. Η αναφορά αυτή θα παραμείνει ανοιχτή, θα αποσταλεί επιστολή στην βουλγαρική κυβέρνηση και στην επιστολή αυτή θα ρωτήσω με τι κάνει η Βουλγαρία με την αποϊδρυματοποίηση και τις βέλτιστες πρακτικές για να ζουν ανεξάρτητα οι άνθρωποι, να μην ε, είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και οι ηλικιωμένοι με, ειδικές, με αναπηρίες να ζουν αξιοπρεπώς. Και τι θα κάνει η Κομισιόν για να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές που συζητήσαμε σήμερα. Επίσης θα πρέπει να είναι βέβαιον ότι και τα κονδύλια θα βοηθήσουν στη μετάβαση τη βουλγαρική κυβέρνηση γιατί συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κόσαφ η Ευρώπη κάνει μια προσπάθεια βοηθάει και η Κομισιόν και θέλουμε να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στη μετάβαση ώστε τα παιδιά να τοποθετούνται σε οικογένειες και να αντιμετωπίζονται σωστά οι αναπηρίες. Θα κρατήσουμε λοιπόν την αναφορά ανοιχτή και θα δούμε τι θα πει και η βουλγαρική κυβέρνηση. Είμαι πεπισμένη ότι η βουλγαρική κυβέρνηση εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είπε και η Κομισιόν και δικαιούται να υποστηριχθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν γράψετε επιστολή στη βουλγαρική κυβέρνηση και στην Κομισιόν είναι σημαντικό να δώσετε σωστό ορισμό της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης. Τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση, γιατί καμιά φορά υπάρχουν παρερμηνίες και αυτές δεν οδηγούν. Βεβαίως, βεβαίως, αυτό θα το κάνουμε. Ωραία, και έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και πάμε στο σημείο 23. Πού είναι η Αντιπρόεδρος? Ε, είμαστε στην αναφορά 145-2019 από τον Ισμέλ Αντώνιο Λόπε Πέρε, Ισπανό πολίτη, εκ μέρου τη οργάνωση Πετών Τελόμπο, μια περιβαλλοντική οργάνωση που ε, ζητάει να εξεταστεί ένα δάνειο που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην εταιρεία Grenalia Biomass Power τη Τεξέιρο στην περιοχή Λακορούνια τη Γαλλικία. Ε, ο κύριο Τζούλιο Μπόλμπι, ε, εκ μέρου τη Κομισιόν, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνοψίσω την ανάλυση μας σχετικά με την αναφορά αυτή. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο αναφέρον εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την ε, βιωσιμότητα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του έργου που είναι μια, ένα σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 50 ΜΒ από βιομάζα. Εξετάσαμε τις πληροφορίες που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις ε, ε, προαπαιτήσεις που θέτει, τις προδιαγραφές που θέτει ε, η ΕΤΕ, ε, δηλαδή πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική κοινωτική νομοθεσία και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ανασώσιμε Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον απαιτείται ε, πιστοποίηση μέσω ε, FSC, DFSC, δηλαδή εθελοντικά συστήματα ε, διαπίστωσης, διαπίστευσης και ότι δεν χρησιμοποιείται στο έργο βιομάζα εισαγόμενη από, από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες του σχετικά με την εφορία ενός τέτοιου σχεδίου χρήσης ε, στερεάς βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά θα θέλαμε να ε, σας πούμε ότι με την ε, αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες που θα ενταχθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021 στις εθνικές νομοθεσίες, η οδηγία αυτή περιλαμβάνει ένα πολύ πιο ενισχυμένο πλαίσιο εφορίας που ε, καλύπτει όλες τις χρήσεις της βιομάζας, περιλαμβανομένων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και περιλαμβάνει ειδικά κριτήρια βιωσιμότητας για την βιομάζα δασικής προέλευσης κάθε δηλαδή ε, βιομάζα δασικής προέλευσης που χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό τομέα ενέργειας πάνω από κάποιο κατόφλι για μεγάλη κλίμακα δηλαδή σταθμούς παραγωγής πάνω από τα 20 ΜΒ. Αυτό δηλαδή, το, αυτή η μονάδα για την οποία μιλάμε σίγουρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο κριτήριο αηφορίας. Ε, εξετάσαμε λοιπόν ε, τα παράπονα και τις ανησυχίες που εκφράζονται και θεωρούμε ότι η ε, φορεία της ε, μονάδας αυτής ε, που χρησιμοποιεί βιομάζα θα εξασφαλιστεί μέσω της αναθεωρημένης οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την παρουσίαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ο αναφέρον. Δεν υπάρχει αναφέρον, δεν είναι εδώ αλλά προφανώς ε, θα θέλει εδώ λόγο ο κύριος Κάλεφος, συνάδελφός μας. Ευχαριστώ. Η πρότασή, μας, ε, η πρότασή μου θα ήταν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να προσπαθήσουμε να την διερευνήσουμε κάπως περισσότερο. Κυρίως γιατί βλέπουμε τόσες πολλές αναφορές που σχετίζονται με ε, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν βιομάζα. Άρα υπάρχει ένα συστηματικό πρόβλημα ε, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εμβαθύνουμε τη διαρεύνησή μας γιατί η βιομάζα είναι εξαιρετική σημασία για την... Ε, πολιτική μα για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε τέτοιου είδου εγκαταστάσει και τον τοπικό πληθυσμό που φαίνεται να υπάρχει σε πολλέ περιπτώσει. Η σκέψη μου λοιπόν είναι να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να δείξουμε ε, μεγαλύτερη προσοχή ε, σε θέματα που αφορούν την ε, βιομάζα και τις σχετικές αναφορές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την σημαντική σας η υπόδειξη και ίσως και κατάληξη της σύντομης αυτής της συζήτησής μας. Θα ήθελα κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρότασή σας και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και η απόφασή μας είναι ότι το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Έχουμε την αναφορά υπαριθμών 143 από τον Αλεχάνδρο Μπλάσκο από την Ισπανία εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της ΡΕΑΛ σχετικά με το κλείσιμο και το σφράγισμα και την περιβαλλοντική αποκατάσταση ε, ε, ε, χωματερών που βρίσκονται σε αχρηστία στην, ε, στο Δήμο της Ρεάλ στην Βαλένσια. Πρώτα απ' όλα, ο αναφέρον. Α, δεν είναι εδώ, μάλιστα. Τώρα. Χωσέ Ντίας Τελ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Η αναφορά αυτή μας ήρθε πέρυσι Κοινοποίησαμε το γεγονός στην Περιφερειακή Διοίκηση της Βαλένσια και πήραμε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δύο χωματερές που βρίσκονται σε αχρηστία στην περιοχή αυτή ε, τον Οκτώβριο που μας πέρασε πέρυσι. Στη συνέχεια ενημερώσαμε εδώ την Επιτροπή σας σχετικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα γεγονότα. Υπάρχουν εδώ δύο χωματερές που αναφέρονται στην αναφορά. Ε, για δημοτικά απόβλητα είναι η μία ε, και οι άλλοι για επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Ε, έχουν, έχει σφραγιστεί και, και κλείσει η μία από αυτές τις χωματερές. Υπάρχουν όμως διαρροές ε, και ε, υπάρχει εκπομπή αερίων, πράγμα και γίνεται καύση του αερίου όπως το απαιτεί η νομοθεσία. Ε, η... Ζητήθηκε από το Δήμο της Ρεάλ, όπου βρίσκονται αυτές οι χωματερές, να δώσουν ενημέρωση για το κλείσιμο της εγκατάστασης αυτής. Δυστυχώς ε, έχει καθυστερήσει η ενημέρωση αυτή έχει καθυστερήσει στις ε, υπηρεσίες ε, επιθεώρησης. Φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να επανενεργοποιηθεί αυτή η χωματερή και η Γενεραλιτά, η αρμόδια δηλαδή τοπική αρχή, προχώρησε ε, στο αίτημα αυτό να ανα να αποκατασταθεί η χωματερή αυτή. Τώρα για την άλλη χωματερή, για τα επικίνδυνα απόβλητα, αυτή ήταν κάπως πιο προβληματική. Πρώτα απ' όλα ε, κινήθηκαν δύο πειθαρχικέ διαδικασίες. Μία το 2004 για το σφράγισμα και την αποκατάσταση της ε, τοποθεσίας αυτής. Ο ιδιοκτήτης τότε Τη εγκατάσταση. ε, ενημέρωσε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εργασίες γιατί και πάλι ο Δήμος της Ρεάλ δεν είχε δώσει την έγκριση του. Βλέπουμε δύο παίκτε λοιπόν εδώ. από τη μια ο Δήμος και από την άλλη η Περιφέρεια που έχει πάρει την πρωτοβουλία για να ζητήσει συμμόρφωση με την ομοθέσια Και πάλι το 2013 κινήθηκε μια άλλη πειθαρχική διαδικασία. Αυτή τη φορά ξεκίνησε από από την υδρογραφική ε, επιθεώρηση με το φόβο ότι τα υλικά που περιέχονται στην χωματερή μπορεί να είναι σε επαφή με κοντινά εκεί ποτάμια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι δύο πειθαρχικές διαδικασίες δεν έδωσαν αποτελέσματα και στη συνέχεια η Γενεραλιτάτ και πάλι δηλαδή οι περιφερειακές αρχές μας ενημέρωσαν ότι οι σχετικές εργασίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και για τους λόγους αυτούς ε, συνεχίζουν να προσπαθούν να συντονίσουν όλους τους εμπλεκόμενους ε, σε αυτή την υπόθεση. Αυτά προς το παρόν έχει η Κομισιόν να ε, σας αναφέρει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ενημέρωση. Και τώρα η κυρία ε, Πινέρο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Κομισιόν για την ενημέρωση που μας έδωσε και για το έργο τους. Εγώ μιλώ για τη σοσιαλιστική ομάδα, είμαι από τη Βαλένθια και ξέρω το πρόβλημα των τοπικών αρχών στη ΡΕΑΛ. Οι δύο χωματερές ήταν πρόβλημα για χρόνια. Ε, συμφωνούμε απόλυτα με τις ανησυχίες του αναφέροντος και πολλών άλλων που ζουν στην περιοχή Ρεάλ. Και εδώ και μια δεκαετία ζητούν την στεγανοποίηση και αποκατάσταση αυτών των χωματερών. Εν τω μεταξύ περνάει ο χρόνος και πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτό που είναι πρωτόγνωρο είναι ότι ο ανεφέρον, ο Αλεχάνδρο Μπλάσκο Σάντσεθ, ήταν δήμαρχος για πολλά χρόνια αυτής ε, της πόλης και εκείνος δυσκόλεψε το έργο σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε το 2012 όταν ο αναφέρον ήταν ε, δήμαρχος η υπηρεσία περιβαλλοντικών ελέγχων που είναι περιφερειακή αρμοδιότητα δεν έλαβε καμία απάντηση σχετικά με τη στεγανοποίηση και αποκατάσταση αυτών των πρώην χωματερών, ενώ θα έπρεπε να γίνει αυτό. Και επίσης ανησυχούμε διότι το 2006 και το 2007 η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έκανε δεκτές άδειες για τη στεγανοποίηση και αποκατάσταση των, της τοξικής χωματέρης. Και φαίνεται ότι δεν έγινε κανένα έργο κατόπιν τούτου. Οπότε ανησυχούμε, διότι το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί λόγω της ρήπανσης ε, των υδάτων στην περιοχή και της γενικότερης ρήπανσης. Και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι τοπικοί άρχοντες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, τόσο ώστε να ε, συμμορφωθούν προς το περιβαλλοντικό δίκαιο. Μου λέγουν επίσης ότι η τωρινή τοπική αυτοδιοίκηση που είναι από άλλο πολιτικό κόμμα έχει εκδώσει τις άδειες οπότε είναι δυνατόν τις επόμενες εβδομάδες να στεγανοποιηθεί η τοξική χωματερή και υπάρχει και πρόβλεψη αναδάσωσης της περιοχής εκεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και να γίνει ένα φωτοβολταϊκό εργοστάσιο, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός. Ε, η ομάδα μου ζητεί να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες σωστά. Και πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε ότι έγινε το έργο. Η Επιτροπή αυτή μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως και η επιθεώρηση από την κοινότητα της Βαλένθια. Μέχρι να γίνει δουλειά πρέπει η αναφορά να μείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκοτικάνεφ, Κάνεφ. Να υποστηρίξω και εγώ τον συνάδελφο και να πω ότι φαίνεται προφανές ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Α, δεν έχουμε, πολλές πληροφορίες δεν έχουμε για να αποφασίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς ζητεί το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και θα στείλουμε και στην Generalitat Βαλεντιάνα μία επιστολή για να ε, παρακολουθήσουν την κατάσταση και να μας ενημερώσουν για τη διαδικασία αποκατάστασης αυτών των χωματερών. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τόπος και χρόνος της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Πέτει 16 Μαρτίου 2020 να αρχίσουμε στις 3 το απόγευμα και να τελειώσουμε στις 6 και μισή το απόγευμα και την επόμενη μέρα στις 17 Μαρτίου να αρχίσουμε το πρωί στις 9 μέχρι τις 12.30 και θα συνεχίσουμε το απόγευμα. Θα αρχίσουμε 2.30 και ως ήθιστε θα τελειώσουμε στις 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις νομίζω. Ευχαριστώ για την ε, ενεργό σας απουσία και καλή σας όρεξη.